colleagues, Συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση. Ζήτω συγγνώμη για την καθυστέρηση. Ζητώ συγγνώμη και ευχαριστώ τους συναδέλφους που ήταν εδώ το πρωί. Είχαμε πολύ δύσκολη συνεδρίαση σήμερα το πρωί. Κάποιοι συνάδελφοι έπρεπε να αποχωρήσουν και κάποιοι νομίζω εξαντλήθηκαν. Σας ζητώ συγγνώμη, πάντως είναι πολύ σημαντικό το θέμα που έχουμε τώρα και ευχαριστώ τους συναδέλφους που είναι εδώ για αυτό το θέμα. Πρόκειται για τη συνέχεια που πρέπει να δοθεί στη διακήρυξη της Νέας Υόρκης και χαίρομαι που βρίσκεται εδώ η κυρία Κνούτσεν ε, και πρόκειται για ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το Παγκόσμιο Σύμφωνο για την ασφαλή, ομαλή και νόμιμη μετανάστευση. Um, και να σας δώσω λίγες εξηγήσεις. Ε, πρόκειται για παρουσίαση της ε, Συμβολής Ευρωπαϊκής Ένωσης σε έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ σχετικά με το Παγκόσμιο Σύμφωνο για την Ασφαλή Ομαλή και Νόμιμη Μετανάστευση. περισσότεροι από εσά θα γνωρίζουν ότι είναι θέμα με το οποίο έχει ασχοληθεί η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική ε, Δράση και ο ΙΕΣ στις 19 Σεπτεμβρίου οργάνωσε διάσκεψη κορυφή ε, στη Νέα Υόρκη ε, για τα θέματα μετανάστευση. Υιοθετήθηκε ψήφισμα για καλύτερη ανταπόκριση τη διεθνούς κοινότητα και το Κοινοβούλιο ήταν παρόν με αντιπροσωπεία ad hoc τριών μελών τη επιτροπή ΛΥΠΕ, την κυρία Βίξτρομ. την κυρία Γκράφιν ε, Τον Χόνστιν και την κυρία Ριστάν. Και η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ ως αποτέλεσμα αυτής ε, της ε, συμμετοχής και είχαμε και στο παρελθόν συζήτηση με την κυρία Κνούτσεν, επειδή παρακολουθούμε την διαδικασία αυτή. έχει τη σημερινή συζήτηση. Ακούσαμε τον Γενάρη πρώτη φορά την κυρία Κνούτσεν σχετικά με τη συνέχεια που πρέπει να δοθεί στη διακήρυξη και δύο κοινέ προσκλήσεις από την ΛΥΜΠΕ και την ΑΦΕΤ εστάλησαν ε, στον ε, υπατορμοστή για τους πρόσφυγες ε, και στον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης. Έτσι δεν είναι, ναι. Έχουν σταλεί λοιπόν αυτές οι προσκλήσεις. Τώρα όμως με πολύ χαρά θα δώσω το λόγο στην κυρία Κνούτσεν για να ακούσουμε τους δικούς της προβληματισμούς σχετικά με την διαδικασία αυτή. Χαίρομαι πάρα πολύ που ε, έχει αποδεχθεί την ε, πρόσκλησή μας. Ε, Λότε, ευχαριστώ πάρα πολύ που βρίσκεσαι εδώ. Σου δίνω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση να σας δώσω πληροφορίες σχετικά με το σύμφωνο για την μετανάστευση και τη σχετική διαδικασία. Ε, είπατε ότι θα προσκαλέσετε τον κύριο Γκράντι και την ε, κυρία Σουίφτα αρχές του 2018. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη μέση της ε, διαδικασίας. Εάν λοιπόν οργανώσετε μια τέτοια ανταλλαγή απόψεων αρχές του 2018 θα είναι πολύ καλή στιγμή εν ώψη του σχεδίου του κειμένου που θα τεθεί επιτάπητος. Πριν από ένα χρόνο λοιπόν με την διακήρυξη της Νέας Υόρκης ε, ξεκίνησε η διαδικασία, 193 ε, χώρες ε, το προσπέγραψαν και η διαδικασία προβλέπεται να ολοκληρωθεί του χρόνου τον Σεπτέμβριο. Δηλαδή βρισκόμαστε ακριβώ στα μέσα του δρόμου και ίσω γι' αυτό δεν συζητήθηκε πολύ η μετανάστευση στην Ούγκα, στην Γενική Συνέλευση. Ε, αλλά ο κύριος Κουτιέρης, ο κύριος Λάιτσακ, ο κύριος Κράντι, ο κύριος Σουίν και ε, ο κύριος Άρβα που επίσης έχει επισκεφτεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, συμμετείχαν σε μια εκδήλωση που στόχο είχε να δείξει ότι βρισκόμαστε στα μέσα μιας διαδικασίας. Χρειάζεται να διατηρήσουμε την ορμή διότι υπάρχει βούληση, υπάρχει φιλοδοξία να προχωρήσουμε και να διασφαλίσουμε το σύμφωνο να είναι ένα καλό τελικό προϊόν με τη συμμετοχή όσο γίνεται περισσότερων χωρών. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικά όλα αυτά και χαίρομαι πάρα πολύ που ενδιαφέρεστε για το θέμα. Ε, έχει να κάνει με τη μετανάστευση, αλλά πρέπει να τονίσουμε ότι επειδή είναι διακήρυξη του ΟΗΕ, έχει να κάνει και με ε, την πολυμερή διαδικασία την οποία θέλουμε να στηρίξουμε. Δηλαδή, στήριξη του ΟΗΕ, του κυρίου Κουτιέρες, με ένα ε, ισχυρό ε, διεθνές σύστημα το οποίο να βασίζεται σε κανόνες. Αυτό λοιπόν είναι το γενικότερο πλαίσιο. Αυτή τη στιγμή φτάνουμε στα τέλη της διαδικασίας διαβούλευσης. Δεν ξέρω εάν ευρωβουλευτές έχουν συμμετάσχει στις ε, θεματικές διαβουλεύσεις που πραγματοποιήθηκαν ε, στη Νέα Υόρκη και την Βιέννη πάνω σε μια σειρά θεμάτων. Δεν χρειάζεται να μπω σε λεπτομέρειες, απλά να σας πω ότι το τελευταίο εξάμεινο είχαμε μια ε, πολύ πλούσια διαδικασία διαβούλευσης και η Λίζα Άρμπορ που είναι Γενική Γραμματέας για το θέμα της μετανάστευσης μαζί με τον Ελβετό και Μεξικανό διαμεσολαβητή ε, είχαν μια πολύ επικοδομητική διαδικασία πολύπλοκη, διότι είχαμε ε, θεματικές διαβουλεύσεις που κάλυπταν μια σειρά θεμάτων ε, από ανθρώπινα δικαιώματα μέχρι αντιξιακή βοήθεια και έγιναν και περιφερειακές διαβουλεύσεις. Έχουν όμως ε, ασχοληθεί πολύ με θέματα μετανάστευσης και έχουν επιτρέψει σε διάφορες ομάδες συμφερόντων από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και ε, κράτη-μέλη του ΟΗΕ και την κοινωνία των πολιτών να συμμετάσχουν σε αυτές τις συναντήσεις διαβουλεύσεων. Έχουν συγκεντρώσει λοιπόν πάρα πολλές πληροφορίες. που έχουν συγκεντρωθεί για πολύ συγκεκριμένο στόχο. Έχουν συγκεντρώσει λοιπόν πληροφορίες, ε, στατιστικά στοιχεία με στόχο την προετοιμασία της διαδικασίας ε, διαπραγμάτευσης. Ε, για κάθε διαβούλευση λοιπόν υπάρχει πολύ πλούσιο υλικό στην ιστοσελίδα για το σύμφωνο όπου συνοψίζονται οι διάφορες διαβουλεύσεις που πραγματοποιήθηκαν. Στο τέλος της διαδικασίας αυτής λοιπόν τώρα πια προετοιμαζόμαστε για την προπαρασκευαστική διάσκεψη στο Μεξικό που συνδιοργανώνουν ε, ο Ελβετός και ο Μεξικανός ε, συνδιαμεσολαβητής. Στόχος είναι να έχουμε μια ευρύτερη συζήτηση, να έχουμε το απόσταγμα όλων των διαβουλεύσεων, να δούμε πού βρισκόμαστε και Πού θέλουμε να φτάσουμε με το σύμφωνο και να έχουμε συζητήσεις, να συμπληρώσουμε τα κενά και να εξετάσουμε τι συνέχεια θα πρέπει να δοθεί στην διακήρυξη εν ευθέτω χρόνο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρεται ε, ρητά ως ε, συμμετέχον στο Μεξικό και Το Μεξικό ε, επισημαίνει την σημασία της ενεργού συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κάτι που σκοπεύουμε να κάνουμε. Στο Μεξικό λοιπόν θα είμαστε τρεις μέρες και ίσως θα έπρεπε να ε, αναφέρω πριν με ρωτήσει κανείς ότι υπάρχει δυνατότητα και για Ευρωπουλευτές να συμμετάσχουν στην ε, ε, στους, ε, θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν και οι ευρωβουλευτές. Οι δύο πρόεδροι θα προσπαθήσουν ε, να συνθέσουν όλα όσα θα τεθούν εκείνες τις τρεις μέρες σε μια σειρά από συζητήσεις με πάνελ. Και αυτά θα αποτελέσουν τη βάση για το σχέδιο μηδέν το αρχικό σχέδιο το οποίο θα είναι βάση των διαπραγματεύσεων αρχές Φεβρουαρίου και κατόπιν θα ακολουθήσουν έξι μήνες εντατικών διαπραγματεύσεων, ε, ουσιαστικά ένα τριήμερο το μήνα. Αυτά σχετικά με το θέμα αυτό. Ε, σήμερα έχουμε διανύμει και ζητώ συγγνώμη που το διανύμαμε τόσο ε, αργά, με τόση καθυστέρηση. Έχουμε διανύμει όμως την συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Λουίς Άρμπερ ε, συνοδεύει το σύνολο της διαδικασίας, ε, συμμετέχει μαζί με τους συνδιαμεσολαβητές και το καθήκον της ε, είναι να υποβάλει έκθεση από πλευράς του Γενικού Γραμματέα, του κυρίου Γκουτιέρες, η οποία μάλλον θα δημοσιευτεί αρχές Δεκεμβρίου πριν τα Χριστούγεννα, η οποία θα καλύπτει το σύνολο της διαδικασίας και χωρίς να θέλω να προδικάσω τις ε, πράξεις της, ε, μάλλον ε, θα υποδείξει το δρόμο για μια στρατηγική, για ένα μελλοντικό όραμα για την μετανάστευση που θα ξεκολλάει από τις προκαταλήψεις του παρελθόντος. Το έγγραφο αυτό θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους συνδιαμεσολαβητές ως βάση για το λεγόμενο μηδενικό έγγραφο. Η όλη διαδικασία είναι διαφανής και συμμετοχική. Θα συμμετέχουν οι χώρες μέλη του ΟΗΕ και η κοινωνία των πολιτών. Η Λουίζα Άρπορ λοιπόν ζήτησε ε, συνεισφορές ε, από ευρία γκάμα χωρών ε, και άλλων παραγόντων. Ρωτάει δηλαδή τις διάφορες χώρες τι θεωρούν ότι θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στο σύμφωνο. Εμείς λοιπόν ε, έχουμε ε, υποβάλει τη συνοσφαρά μας την οποία έχουμε διανύμει. Αποτελεί κατευθυντήρια γραμμή, τίποτα παραπάνω. Είναι κάτι που έχουμε συζητήσει με τα κράτη-μέλη. Εάν θέλουμε να έχει επιτυχή έκβαση αυτή η διαδικασία, είναι πάρα πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι ενωμένη. Ενώ λοιπόν αυτή η συνεισφορά δεν ε, εμποδίζει τα κράτη-μέλη να υποβάλουν δικές τους μεμονωμένες συνεισφορές, ε, ουσιαστικά σκιαγραφεί αυτά που θέλουμε να πετύχουμε. Κάποιες παρατηρήσεις σχετικά. Έχουμε υποβάλει κάποιε ιδέε ε, υπό τέσσερι διαφορετικού τίτλου. Σε τίποτα δεν θα σα εκπλήξει. Ακολουθούν τη διακήρυξη τη Νέα Υόρκη, που ήταν ένα πολύ φιλόδοξο έγγραφο και νομίζω ότι υπάρχει γενική συνένεση ότι μάλλον περιέχει όλα τα θέματα στα οποία θα πρέπει να εμβαθύνουμε και τα οποία θα πρέπει να αναπτύξουμε στη συνέχεια. Όσον αφορά λοιπόν το γενικό αφήγημα, ε, καταρχάς ε, θέτουμε το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, των μεταναστών με ιδιαίτερο επίκεντρο την προστασία και βοήθεια ιδιαίτερα ευάλωτων μεταναστών και παιδιών, καθώς και το θέμα της ισότητας των δύο φύλων. Το δεύτερο θέμα έχει να κάνει με τις αιτίες της μετανάστευσης Εξετάζουμε λοιπόν τους παράγοντες που οδηγούν τους ανθρώπους στη μετανάστευση. Είτε οι αιτίες αυτές ε, είναι ανθρωπογενείς, ε, πολιτικές, ε, εγχώριες εξελίξεις, είτε έχουν να κάνουν με φυσικές καταστροφές. Έτσι λοιπόν ασχολούμαστε με τις αιτίες της μετανάστευσης και εξετάζουμε θέματα όπως είναι η πρόληψη συγκρούσεων ε, η... και η ανθεκτικότητα απέναντι σε αυτές. Η τρίτη ομάδα θεμάτων έχει να κάνει με την ε, μετανάστευση και την ε, ανάπτυξη. Είναι σημαντικό να βλέπουμε τη μετανάστευση μέσα από τον φακό της ανάπτυξης. Η μετανάστευση λοιπόν μπορεί να ενισχύσει την ανάπτυξη και αντιστρόφως. Εξετάζουμε λοιπόν εδώ τρόπους σε συνεργασίες με χώρες προέλευσης ή διέλευσης καθώς και χώρες προορισμού των μεταναστών. Ε, εξετάζουμε τις διάφορες ε, αναπτυξιακές πτυχές όπως είναι ε, τα εμβάσματα που στέλνουν οι μετανάστες στις πατρίδες τους κλπ. Η τέταρτη ομάδα θεμάτων έχει να κάνει με την διακυβέρνηση. Πιστεύουμε ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα. Έχουμε τον νότιο άξονα αλλά και τον ε, άξονα βορρά-νότου ε, στη μετανάστευση. Σκοπός είναι λοιπόν ε, να μπορούμε να έχουμε ασφαλή, ομαλή μετανάστευση. Θίγουμε λοιπόν εδώ μία σειρά θεμάτων που έχουν να κάνουν με την ε, τεχνική βοήθεια και υποστήριξη, ε, συνεργασία, εθελοντική επιστροφή με αυστηρό σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πέμπτη ομάδα θεμάτων έχει να κάνει με την αντιμετώπιση της ε, ε, παράνομης μετανάστευσης, την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και έχει να κάνει με το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τις χώρες ε, να παρεμποδίζουν τις ε, ενέργειες των διακινητών. Η έκτη ομάδα θεμάτων έχει να κάνει με τις νόμιμες οδούς μετανάστευσης και έχει να κάνει με το πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ευκαιρίες απασχόλησης, κινητικότητα εργαζομένων και να ενισχύσουμε το δυναμικό στις χώρες υποδοχής. Όπως και να έχει, αυτές είναι οι ομάδες θεμάτων, ε, πιθανότατα να ομαδοποιηθούν διαφορετικά στο τελικό σύμφωνο. και στο Μεξικό και στις διαπραγματεύσεις στη συνέχεια. Σημαντικό ρόλο θα παίξει ο μηχανισμός ε, για τη συνέχεια που θα δοθεί, το follow-up mechanism. Ε, δεν θέλουμε να έχουμε... ένα μεμονωμένο περιστατικό ε, θέλουμε να έχουμε συνεχή παρακολούθηση και επίσης ε, αυτό που συζητιέται είναι να έχουμε ένα μη δεσμευτικό έγγραφο, ένα όχι νομικό έγγραφο, να έχουμε έναν μηχανισμό παρακολούθησης που να μην οδηγεί σε νέες δομές και αυτό αποτελεί κόκκινη γραμμή στις διαπραγματεύσεις, αλλά έναν τρόπο συνεργασίας με χώρες σε όλο τον κόσμο για να διασφαλίσουμε την ε, συνέχεια. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να γίνει αυτό, υπάρχουν διάφορα φόρουμ στα οποία μπορεί να γίνει αυτό. Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης ε, σίγουρα μπορεί να παίξει ρόλο και μπορεί να υπάρχουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι όπως είναι ε, το Παγκόσμιο Φόρουμ για την Μετανάστευση και Ανάπτυξη, το Φόρουμ τη Ούγκα. Σίγουρα όμω θα πρέπει να αποφύγουμε τη δημιουργία νέων δομών και επικάλυψη δομών και εργασιών θα πρέπει να εξετάσουμε τι θέλουμε να κάνει ο μηχανισμός ε, αναθεώρησης, ο μηχανισμός παρακολούθησης. θα πρέπει να εξετάσουμε τους ε, στόχους μας ε, και να δούμε πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε την συνεισφορά όσο γίνεται περισσότερον. Ενώ αυτή η διαδικασία βασίζεται σε πολλές διαφορετικές ομάδες συμφερόντων, ουσιαστικά πρόκειται για κυβερνητική προσέγγιση και Ε, μπορούμε να πετύχουμε καλό και βιώσιμο αποτέλεσμα αν έχουμε ευρείες επαφές. Πρόκειται δηλαδή για τμήμα μιας μακροπρόθεσμης προσπάθειας ε, και από την Αφρική, τις Αραβικές χώρες, ε, την Ασία θα πρέπει όλοι να συμμετάσχουν αν θέλουμε να έχουμε μια διαρκή διαδικασία. Πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε μια κατάσταση από την οποία να κερδίζουν όλοι και να περιέχονται θέματα ενδιαφέροντος ε, για όλους. Επίσης θέλουμε ένα μη δεσμευτικό πλαίσιο το οποίο να επιτρέπει κάποιο βαθμό ευελιξίας διότι η μετανάστευση είναι ένα διαρκές φαινόμενο. Χρειαζόμαστε όμως ένα πλαίσιο που να έχει αρκετή ευελιξία ώστε να διαρκέσει και να μπορεί να λάβει υπόψη μελλοντικέ εξελίξεις, ώστε να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε στις μελλοντικέ προκλήσεις. Αυτά λοιπόν γενικά και εάν, επανέλθουμε, εάν επανέλθετε στο θέμα αρχές Ιανουαρίου θα γνωρίζουμε περισσότερο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Uh, Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Κνούτσεν. Έχουμε το input paper της Ευρωπαϊκής Ένωσης το αναλύσαμε, ακούσατε την ανάλυση. Όποιοι δεν ήσασταν από την αρχή, εγώ είπα συγκεκριμένα για τη Λίμπε, την Άφετ και την ΤΕΒΕ Τι έχουμε εμείς κάνει για τη διαγεξιάση ορκής και τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Και θα έχουμε σε αρχές του χρόνου κάποιο input και ήταν πολύ χρήσιμο να ακούσουμε την κυρία Κνούτσεν και την ανάλυση της. Υπάρχουν συνάδελφοι που θέλουν το λόγο. Η Έλλη Στάιν ήταν στη Νέα Υόρκη. Ας ξεκινήσει η Έλλη λοιπόν. Σας ευχαριστώ Κλοντ. Να περίμενα να βάλεις τα ακουστικά σου. Σας ευχαριστώ που είστε πάλι μαζί μας και μας δώσατε πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες για το πώς προχωρούν οι διάφορες διαδικασίες και τι συνέχεια δίνεται. Θα θυμάστε ίσως με άλλες συναδέλφους, ήμουνα στην αντιπροσωπεία που <coughs> συμμετείχε στην ε, διάσκεψη κορυφής που έλαβε υπόψη τη σημασία σε μια ιδιαίτερη διεθνή περίσταση. Νομίζω πως είναι καλό να προχωρήσουμε και ίσως και να έχουμε περιμένει και υπερβολικά πολύ και να σας πω μάλιστα ότι μόλις σήμερα το πρωί η Επιτροπή μας έκανε μια πολύ σημαντική ψηφοφορία για την καρδιά του συστήματος ασύλου της Ευρώπης, το Δουβλίνο δηλαδή, θέλησε να δώσει δώσει ένα μήνυμα μοιρασιά τη ευθύνη όσον αφορά την υποδοχή. Είναι μια θέση του Ευρωκοινοβουλίου πολύ χρήσιμη για τη συζήτηση που γίνεται και μάλιστα μετά την διάσκεψη κορυφή της Νέας Υόρκη, όπου δηλαδή ακριβώς το ίδιο ζήτημα μιας δίκαιης μοιρασιά, ευθυνών τίθεται όχι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο ακριβώ, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο, γνωρίζοντα πολύ καλά ότι το 86% των εκδιοχθέντων σε ολόκληρο τον κόσμο ε, φιλοξενούνται σε χώρε αναπτυσσόμενες. Αυτό σημαίνει πω οι πιο φτωχέ χώρε είναι αυτέ που καταβάλουν τις ε, πιο μεγάλε προσπάθειε όσον αφορά την προσπάθεια υποδοχή Γι' αυτό θα πρέπει πολύ να προβληματιστούμε. Ακριβώς το σημερινό αποτέλεσμα μας καθιστά πιο αξιόπιστο όταν είμαστε στη Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων της Νέας Υόρκη και μιλάμε για μεγαλύτερη και καλύτερη μοιρασιά των ευθυνών σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα συνεχίσουμε λοιπόν από αυτή την, από αυτή την Επιτροπή αλλά και εγώ προσωπικά να παρακολουθούμε τις εξελίξεις για να δούμε ε, προς ποια κατεύθυνση προχωράμε ευχαριστώ και ίσως και χάρη στην εργασία για το Παγκόσμιο Σύμφωνο να καταφέρουμε να υπάρξει μεγαλύτερη δέσμευση από πλευρά του πιο πλούσιου κομματιού του κόσμου όταν πρόκειται για την περίθαλψη των όσων το χρειάζονται. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να προσθέσω σε σχέση με αυτά που είπε η Έλλη. Για το πρωί πράγματι η πλειοψηφία ήταν υπέρ του Δουβλίνου αλλά στο πλαίσιο της ανάλυσης. Νομίζω θα βοηθήσει αυτό το εγγράφο όλο το πακέτο για το άσυλο. Είναι καιρός να δούμε πλέον κάποια μετακίνηση και ελπίζω και εμείς να μπορέσουμε πιο συγκεκριμένα και με το Δουβλινό ως Ευρωπαϊκή Ένωση να διαδραματίσουμε το ρόλο μας. Θα ήθελα λοιπόν ε, αυτό να υποθεί. Η Σεσίλ τώρα έχει το λόγο και έγκυε. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ, Κλόντ. Σε ευχαριστώ και εγώ την, ε, την ε, ομιλήτρια και τη συγχαίρω για το τελικό αποτέλεσμα αυτού του εγγράφου που το βρίσκω ιδιαίτερα διορατικό. Εγώ επέστρεψα σήμερα το πρωί από μια πολύ σημαντική αποστολή στην Ιγυρία. Έφτασα λοιπόν σήμερα το πρωί κατευθείαν για να λάβω μέρος στις εργασίες της Επιτροπής αλλά και για να μπορέσω να προσφέρω μια συμβολή των όσων προέρχονται άμεσα από την περιοχή. Εγώ και ο συνάδελφο Λόπες πήγαμε στην Ιγυρία σε μια αποστολή να δούμε την οικοδόμηση δυνατοτήτων για το Κοινοβούλιο και τη Γερουσία. Θελήσαμε να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε και να επιμείνουμε για το Κοινοβούλιο, για το ρόλο ενό Κοινοβουλίου και το ρόλο των βουλευτών που δεν ε, πρέπει να είναι που και που, αλλά να είναι διαρκής και σταθερός, μόνιμος. Μάλιστα, μια διακυβέρνηση πολυεπίπεδη ε, είναι η καλύτερη και πιστεύω σε όλα αυτά ο ρόλος του βουλευτή θα πρέπει να είναι κεντρικός και στην Ιγυρία ε, μιλήσαμε λοιπόν για το ρόλο του βουλευτή και την ενίσχυση αυτού αλλά ε, το κρίσιμο θέμα είναι ότι θα υπάρξει ένα δημογραφικό, μια δημογραφική έκρηξη που θα πρέπει να μας οδηγήσει να σκεφτούμε ποιε είναι τα βαθύτερα αίτια. Δεν αρκεί να επιτιθέμεθα και να κατηγορούμε χώρες, αλλά να δίνουμε συγκεκριμένες απαντήσεις γενικές, προσπαθούμε να διαχειριστούμε με υπεύθυνο τρόπο την κατάσταση. Μιλώ λοιπόν ε, για την τρομοκρατία. Ξέρουμε πολύ καλά το βάρος της τρομοκρατίας. Ε, θα πρέπει να μιλήσουμε για τη σύνδεση μεταξύ μετανάστευσης και κινητικότητας, δυνάμιμες ε, διάβλους για τις οποίες μιλήσαμε και για τις οποίες, μιλήσατε και τι οποίε συζητάμε, αλλά και το θέμα της κλιματικής αλλαγής που ήταν και αντικείμενο μιας ε, ε, ε, ισομερού συνέλευσης που διεξήχθη στο Βανουάτου μάλιστα και μας έδωσαν αφού ανέλησαν το έγγραφο της δήλωσης της Νέας Υόρκης, την εξετάσαμε ολόκληρη, το ψήφισμα που εσείς μας παρουσιάσατε και έκαναν έτοιμα να εισαχθεί και να περιλαμβάνεται εντόνως και η φωνή του κλιματικού πρόσφυγα. Σκεφτείτε ότι σε 20, 50, 30 χρονια 30-50 χρόνια αυτοί οι άνθρωποι δεν θα έχουν πάλι πάνω που να πάνε. Και συμφωνώ με τα όσα έλεγε η συνάδελφος Έλλης Λάιν για τις κοινέ ευθύνε. Αυτό θα πρέπει να γίνει και σε νομικό επίπεδο, νομοθετικό επίπεδο. Δηλαδή τα κρατημέλη όχι μόνο να πούνε ναι απλά συμμεριζόμαστε τις ευθύνε, αλλά να γίνουν και νομοθετικές προτάσεις γιατί δεν υπάρχει κάτι δεσμευτικό. Πρέπει εμείς να το κατοστήσουμε ε, υποχρεωτικό με συγκεκριμένες νομοθετικές πράξεις. Τέλος, Θέλω να κάνω μια έκκληση, γιατί από τότε που έγινε η δήλωση της Νέας Ιάρκης, το παρακολουθώ μέχρι σήμερα ε, και προσπαθώ να το εφαρμόσω και να το περάσω σε όλα τα απαραίτητα όργανα και θα ήθελα να συνεχιστεί αυτή η εμπειρία φτάνοντας και στο Μεξικό. Χράζω και τη βούλησή μου να μπορέσω να συνεχίσω αυτή την πορεία γιατί ακριβώς σήμερα χρειάζεται μια σφαιρική προσέγγιση. το σημειώνουμε, Σεσίλ. Μάλιστα. Κύριε Σαρτζεντίνη, Τζούντιθ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μελέτησα το input αυτό για το Σεπτέμβριο και Ουσιαστικά τι κάνουμε, βάζουμε στα τετραγωνίδια, τι κάνουμε και λέμε ναι, ε, βασικές υπηρεσίες, δημοκρατία, μετανάστες, κλιματική αλλαγή, θετική συμβολή των μεταναστών, ο ρόλος της διασποράς, ε, κοινή ευθύνη, επιστροφές, ε, ένταξη, κοινωνική συνοχή και πρόθεση κάποιων νόμιμων διαδρόμων. Α, ναι, ουσιαστικά τσεκάραμε τα τετραγωνίδια μόνο, παρότι είναι λογική ω προσέγγιση αυτή. Εμεί από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση λέμε ότι δεν θα πρέπει να είναι δεσμευτικά νομικώς δεσμευτική διαδικασία θα πρέπει να είναι μια υπεύθυνη διαδικασία στο πλαίσιο των ήδη υφιστάμενων βημάτων συζήτηση στο ΙΕ, να μην δημιουργηθούν νέες δομές και δι τα κράτη-μέλη να χρειαστεί να καταβάλουν περισσότερα χρήματα αλλά δεν είμαι βέβαιο ότι καταλαβαίνω ποια είναι η προστιθέμενη αξία αυτής της διαδικασίας αν ακολουθήσουμε αυτή την προσέγγιση. Και πώς αυτό θα το συνδυάσουμε με τις δραστηριότητες που αναλαμβάνουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλώ για την πολιτική ε, αντιμετώπιση της μεταναστευτικής προσφυγικής ε, κρίσης. Ναι, για τους νόμους διάβρος να μιλήσουμε, αλλά δεν γίνεται κάτι από ευρωπαϊκής πλευρά τώρα ή τα βασικά αίτια της μετανάστευσης. Αν δείτε τι γίνεται με το Ευρωπαϊκό Καταπίστημα για την Αφρική, θα δείτε ότι στα τέλη του 2016 και μέχρι τώρα το 2017 τα χρήματα έχουν φύγει από τις λιγότερο ανεπτυγμένες προς τις ε, χώρες μεσαίου εισοδήματος και και χρήματα φεύγουν από τις προσπάθειες ή προγράμματα καταπολέμησης τη φτώχεια προ τα προγράμματα ελέγχου των συνόρων και τα σχετικά. Η επένδυση πόρων για να πάρουμε ε, τις επιχειρήσεις από νέους στον Ήγηρα. Εντάξει, εγκληματικές είναι αυτές οι ε, δραστηριότητες, αλλά το να φύγουν αυτά τα χρήματα από εκεί δεν βοηθάμε τελικά την καταπολέμηση της μετανάστευσης, των βασικών αιτίων τη μετανάστευση. Το θέμα είναι όχι να μην φύγει ε, ο, ο κόσμος, αλλά να μην φτάσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός είναι ο στόχος μας και δεν ξέρω κατά πόσο αυτή η προσέγγιση είναι υγιεινή. Sorry if, um, you were cut Συγγνώμη που σου έκανα νοήματα, αλλά έπρεπε να έχουμε ολοκληρώσει το θέμα στις 2.30. Παρακαλώ. Όχι, δεν φταίτε εσεί. Εγώ φταίω. Εγώ φταίω ως πρόεδρος, γιατί αργήσαμε να ξεκινήσουμε. Κάνα δύο λεπτά, τελευταία παρέμβαση. Ο Χουάν Λόπεθ. Ευχαριστώ πολύ κύριε πρόεδρε. Δεν μπόρεσα να πάω, ούτε και είχα την πρόθεση άλλωστε να πάω στη Νέα Υόρκη. Άκουσα αυτά που είπε η συνάδελφοι και ιδίω ε, την επίσκεψη στην Ιγυρία Life complained. Και πράγματι έχουμε ένα θέμα με την προσέγγιση για το ποιο θα είναι το μέλλον της πολιτικής που θα ακολουθήσουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαρωτώ με. Πρέπει να έχουμε μια ολιστική προσέγγιση για τη μετανάστευση. Αλλά πού θα εστιάσουμε, στην αρνητική πλευρά, όπως μέχρι τώρα γίνεται. Δηλαδή ότι οι πρόσφυγες είναι ε, κίνδυνος για την ταυτότητα και την ασφάλεια του ευρωπαϊκού κοινωνικού ιστού. Υπάρχει νομίζω το ρητό αίτημα, η ρητή απέτηση να αναθεωρήσουμε την ε, αφήγηση αυτή και να μην ε, τονίζουμε το αρνητικό σκέλος με τις πολιτικές. η διασύνδεση όλων των συμφωνιών με την ικανότητά του να εφαρμόσουν πολιτικές επιστροφής. Αυτό το βλέπουμε, είναι σταθερά στις συνομιλίες που έχουμε με τις χώρες αυτές. Είναι μία ψύχωση με τις επιστροφές και γι' αυτό υπάρχει και αυτή η αρνητική αντίληψη. Συνεχίζουμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το συζητούμε. Θα ήθελα να ξέρω κατά πόσον αυτή η αρνητική προσέγγιση έχει εντοπιστεί και ταυτοποιηθεί ως μέρος του προβλήματος και όχι της λύσης σε διεθνείς ε, διασκέψεις. Σε ευχαριστώ πολύ, Χουάν. Θα σας ξαναδώσω το λόγο, μήπως μπορείτε να απαντήσετε σε αυτά που είπαν ε, η κυρία ε, Σαρτζεντίνη, η οποία ανέφερε και την ε, νόμιμη μετανάστευση. Το Κοινοβούλιο προοδεύει πάνω στο θέμα αυτό και αυτό ανέφερε και η κυρία Σλάιν. Στο έγγραφο αυτό λοιπόν ε, νομίζω ότι λέμε σωστά πράγματα, αλλά ίσως θα έπρεπε να Σημειώσετε ότι σημειώνουμε πρόοδο σε ένα πολύ δύσκολο θέμα. Λέμε στο Συμβούλιο όμως ότι αυτό είναι ένα πιθανό σημείο εκκίνησης. Μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρατάμε ζωντανό το θέμα της νόμιμης μετανάστευσης. Το Κοινοβούλιο δεν σταματάει, όπως άλλωστε είδαμε και σήμερα το πρωί, παρότι είναι πολύ δύσκολο πολιτικά θέμα. Νομίζω λοιπόν ότι σωστό είναι να συμπεριληφθεί και αυτό στο έγγραφο, το οποίο όμως έχει πολύ σωστούς ε, τίτλους ε, και ομάδες θεμάτων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να σας συγχαρώ για τη δουλειά που κάνατε σήμερα το πρωί πάνω στην πρόταση του Δουβλίνου. Σημειώνω αυτά που είπατε και νομίζω ότι αυτό είναι το μήνυμα που μπορούμε να μεταφέρουμε στο Μεξικό θα μπορούσε να συμπεριλαμβάνεται στην δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι προσπαθούμε να πετύχουμε πρόοδο είτε πάνω στο Δουβλίνο είτε στο πλαίσιο πιλωτικών προγραμμάτων στο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για τη Μετανάστευση. Πρέπει λοιπόν και αυτό να το λάβουμε υπόψη μας ως ε, τμήμα μιας ισορροπημένης προσέγγισης. Ε, σημειώνω την ε, παρατήρηση αυτή σχετικά με την ε, αρνητική προσέγγιση. Αυτό που προσπαθούμε να καταφέρουμε μαζί με πολλές ε, χώρες εταίρους μας στην Αφρική είναι ακριβώς αυτό, ότι πρόκειται για εταιρική σχέση και όλη αυτή η διαδικασία βασίζεται στην ολιστική προσέγγιση. Μία ευρεία προσέγγιση ώστε στο τέλος να έχουμε μια κατάσταση από την οποία να κερδίζουν όλοι και να μην ε, επικεντρωθούμε αποκλειστικά στη μετανάστευση, διότι ε, γνωρίζουμε ότι αυτό δεν οδηγεί πάντα στο πιο ε, ισορροπημένο και ολιστικό αποτέλεσμα. Και χαίρομαι που αναφερθήκατε στην Ιγυρία, διότι είναι πολύ καλό παράδειγμα χώρας όπου θα πρέπει να εξετάσουμε τη συνολική εικόνα. Όχι μόνο είναι η χώρα της Αφρικής με το μεγαλύτερο πληθυσμό, Προσπαθούμε να εξετάσουμε διάφορους τομείς πολιτικής και είναι σημαντική η μετανάστευση. Φυσικά θέλουμε να σώσουμε ζωές ανθρώπων. Έχουμε όμως και την αλλαγή του κλίματος και ε, θέλουμε να επικεντρωθούμε και στις ε, βλαβερές συνέπειες, στις αρνητικές συνέπειες της αλλαγής του κλίματος. Ε, θέλουμε λοιπόν να εξετάσουμε τα συνολικές δέσμες μέτρων για τις χώρες αυτές. Υπάρχουν ε, μέρη της χώρας όπου χρειάζεται επιροχνομοσύνη στην γεωργία ε, για την ε, ανάκτηση των πόρων. Θα πρέπει λοιπόν να διορθώσουμε την ιδέα ότι επικαιρωνόμαστε στις αρνητικές συνέπειες. Πρέπει λοιπόν να έχουμε σωστή διαχείριση για να αποφύγουμε την απώλεια ζώων. Όσον αφορά το θέμα της ε, πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, ε, συμφωνώ απολύτως. Ενώ το σύμφωνο της Νέας Υόρκης θα είναι διακυβερνητικό, νομίζω ότι η συμμετοχή ε, διαφόρων ομάδων συμφερόντων είναι πολύ σημαντική. Άλλωστε ζούμε σε έναν κόσμο όπου χρειαζόμαστε τοπικές αρχές, περιφερειακές αρχές, βουλευτές. Γι' αυτό ακριβώς πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντική η συνεισφορά σας και γι' αυτό λέω ότι υπάρχει δυνατότητα για μέλη του Κοινοβουλίου να συμμετάσχουν στην διάσκεψη στο Μεξικό. Και πολύ ευχαρίστως ε, θα λάβω τα στοιχεία τα σχετικά με την Ιγυρία, διότι θα πρέπει να ταιριάξουμε τις διάφορες ε, διαδικασίες ενημέρωσης, ε, ώστε να αποφεληθούμε όσο γίνεται περισσότερο. Νομίζω ότι έτσι κάλυψα τα τρία βασικά θέματα. Οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ξεκινήσει. Η δική μας συνεισφορά αποτελεί προσπάθεια να φροντίσουμε όλα τα θέματα που μας ανησυχούν τελικά ίσως υπό διαφορετική μορφή και ίσως ε, με διαφορετική ομοδοποίηση να ε, συμπεριλαμβάνονται στη λύση. Είναι λοιπόν καλύτερο να τα αναφέρουμε αυτά ήδη στην αρχή. Όσον αφορά την προστιθέμενη αξία πιστεύω ότι η διαδικασία της Νέας Υόρκης αποτελεί πολύ σημαντικό ποιοτικό βήμα προόδου. Αλλάζει το παιχνίδι. Είναι σημαντικό το ότι θέτουμε τη μετανάστευση στον Διεθνή Χάρτη, ότι στον ΟΗΕ συζητιέται, εκεί θα πρέπει να παραμείνει το θέμα αυτό, διότι έτσι έχει διαφορετικού είδους... Ε, ε, έτσι, έτσι γίνεται ορατό με τελείως διαφορετικό τρόπο και αυτή τη στιγμή είναι σωστό να είναι μη δεσμευτικό ε, για παράδειγμα στην Ούντο και στην έχουμε ε, ακόμα συζητήσεις ε, σχετικά με τη συνέχεια που θα πρέπει να δοθεί. Πρέπει λοιπόν να πούμε ότι ναι μπορούμε να συνεισφέρουμε στη διαδικασία και πρέπει να μάθουμε από τους άλλους. Και εδώ ακριβώς έχετε να παίξετε σημαντικό ρόλο. Ο σκοπός είναι να υπάρχει αυτή η αίσθηση οικείωσης ε, με συμμετοχή 193 χωρών ε, θέλουμε να τονίσουμε την αλληλεγγύη και να έχουμε συλλογική προσπάθεια. Αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ. Και σας ευχαριστώ που σε τακτική βάση έρχεστε εδώ να μας ε, κάνετε τέτοια παρουσίαση. Έκλεισε το μικρόφωνο του Προέδρου. Είμαστε λοιπόν αποφασισμένοι να ε, συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας στο θέμα αυτό. Συγγνώμη ζητάει ο πρόεδρος ε, που κλείνει το μικρόφωνο. Έχουμε λοιπόν αρχές του 2018 κάποιες ε, ε, ενέργειες για τη συνέχεια του θέματος αυτού. Έχουμε τη συνάντηση στο Μεξικό. Μας βοηθάτε και εσείς να συνεχίσουμε την παρακολούθηση. Θα συνεχίσουμε λοιπόν αυτήν την οργανωμένη προσπάθεια και θα σας ε, δούμε για να μας κρατήσετε ενήμερους με τις εξελίξεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ και τους ευρωβουλευτές για τη συζητησή τους στη συζήτηση. Um, τη συνάδελφοι, καθυστερήσαμε λίγο, ζητώ συγγνώμη στο συγγνώμη από τον εισηγητή για έκθεση για την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, τον κύριο Έγγελ, εισηγητή μα για το 2017, λέει ο πρόεδρο, είναι από τα πιο αντιπροσωπευτικά έργα τη Επιτροπή μα για τη έκθεση για την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τι προκλήσει στον τομέα τη προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων όλων όσων διαμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγγνώμη που αργήσαμε να ξεκινήσουμε. Θα δώσω το λόγο στον εισηγητή για την ετήσια έκθεση για την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2016. Φρανκ. Thank you, Claude. Σε ευχαριστώ, Κλοντ. Πέμπτη απόγευμα είναι, δεν περίμενα και γεμάτη αίθουσα. Θα είμαι στον πιο ευέλικτος Θα ήθελα να είχα καθίσει βέβαια να φάω με την ησυχία μου το μεσημέρι, αλλά τέλος πάντων ε, την αρχική μου την παρουσίαση θα την κάνω στα γαλλικά και μετά θα σας απαντήσω στις γλώσσες που θα μου κάνετε ερωτήσει. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το σχέδιο έκθεσης για την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2016, αλλά και το 2015, γιατί καταφέραμε για μια κοφά να συνδέσουμε δύο χρόνια, Θέλω να πω τα εξής, καταρχά τη αρχής. Όσοι ήσασταν ε, παρόντες με τους και και άλλους, όλες οι προηγούμενες εκθέσεις ε, είχαν ένα μακρύ κατάλογο των ανησυχιών μας και των μιλημάτων μας για τον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αναφέρονταν επίσης ε, ε, βελτιώσεις για τα δικαιώματα των γυναικών, των ΛΟΑΔ και ούτω καθεξής. Οι προηγούμενες εκθέσεις, στην αρχή τουλάχιστον, προσπαθούσαν να αναφέρουν, όπως είπα, τις ανησυχίες και δι του εισηγητή, τις προσωπικές ανησυχίες του εισηγητού. Εγώ πιστεύω ότι φέτος θέλουμε να βελτιωθεί αυτή η διαδικασία των αιτησιών εκθέσεων, θα πρέπει να εστιάζουμε σε κάποια βασικά δομικά ζητήματα που μας ανησυχούν. Με πιο συγκεκριμένο τρόπο για τα εκάστοτε έτη. Έξω και δεν ήθελα να τα συμπεριλάβω όλα και σίγουρα όχι να κάνω αυτά τα οποία κάνουν οι άλλες εκθέσεις, όπως Ρωμά. Υπάρχει ειδική έκθεση για αυτούς. Βία κατά των γυναικών, δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, ο πλουραλισμό στα μέσα μα και τα κτλ. Αυτά τα θέματα είτε τώρα, είτε πριν λίγο, είτε σε λίγο, θα είναι αντικείμενο ειδικών εκθέσεων εξού και δεν ήθελα να τα συμπεριλάβω για μια κομφρά στην θεσμική έκθεση για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Με αποτέλεσμα αποφάσισα να μιλήσω για τα δικαιώματα και απ' την άλλη για τα, την ολοκλήρωση και τη μετανάστευση. Για τις δύο αυτές χρονιές, 15 και 16, σε ό,τι αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα, που παραμένουν επίκαιρα. Σίγουρα πρέπει να δούμε το πρόβλημα της μετανάστευσης από την πλευρά ενός ε, δουργούντος κράτους δικαίου για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα εμπιστοσύνης των πολιτών στην Ένωση. Το δεύτερο θέμα, το πρώτο λοιπόν είναι η μετανάστευση και το δεύτερο είναι το κράτος δικαίου. Μιλάμε για την ε, Ουγγαρία και για την Πολωνία. Ε, δεν έχει βελτιωθεί τίποτα. Και όσο και πάει και χειροτερεύει το πράγμα. Οι συνεργάτες μου έχει φτιάξει πολύ ωραία φιλμάκια για την ιωστή εθνική διαβούλευση, για κάτι που δεν υπάρχει, το σχέδιο Σόρος συγκεκριμένα, που παίρνει μια τροπή φρικιαστική. Τέλος πάντων, θα σας τα διαβάσω αυτά τα φιλμάκια, αν τα δείτε κι εσείς ε, για την Ουγγαρία. Και το κράτος δικαίου λοιπόν ε, επίσης ε, γίνεται επιστημονική φαντασία εκεί, αλλά γίνεται και στη Μάλτα. Και νομίζω ότι πραγματικά πρέπει να το σκεφτούμε, πρέπει να αγγίψουμε πάρα πολύ προσεκτικά στα θέματα αυτά του κράτους δικαίου. Πρώτο θέμα λοιπόν κράτος δικαίου, δεύτερο μετανάστευση. Παρά τις προσπάθειες σε πολλά κράτη και τα μέτρα που έχει λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση, παραμένουν τεράστια προβλήματα για την υποδοχή, για την κράτηση, για τους ασυνόδευτους ανηλίκους, για την υγεία, την παιδεία κτλ και έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας. Δεν έχουν τελειώσει τα προβλήματά μας. Και έπειτα έχουμε τη ρητορική μίσος, την Ισλαμοφοβία, την Αφροφοβία και όλη αυτή ε, τη κατάσταση. Όλες τις φοβίες αυτές που οφείλονται και σε έλλειψη πολιτικής βούλησης, Αντίδραση σε αυτές τις φοβίες και άσκησης μιας πραγματικής πολιτικής ένταξης ε, η ρητορική βία ε, θεωρείται πλέον κάτι τετριμένο. Και αυτό έρχεται και συνδέεται με την ψηφιακή επικοινωνία και άλλα. Μας ανησυχούν αυτά. Εγώ έχω εστιάσει συνειδητά, όπως είπα, το σχέδιο έκθεσής μου. Και με βάση τον κανονισμό θεσμικά ξέρουμε ότι πρέπει να είναι ε, σύντομης διάρκειας και είπα ποια είναι τα δύο θέματα, κράτος δικαίου, μετανάστευση, ένταξη. Φαντάζομαι ότι θα προσθεθούν κάποια νέα στοιχεία, θα τα προσθέσω και εγώ και άλλοι συνάδελφοι φαντάζομαι θα καταθέσουν τροπολογίες καλοδεχούμενες. Απλά απευθύνω μια έκκληση, την ίδια έκανε και στους κοιότητες εισηγητές. Να προσπαθήσουμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο συνοπτικοί και να μην καταθέσουμε χίλιες τροπολογίες να έχει έκθεση 50 σελίδες και όχι 4, όπως γίνεται κάθε χρόνο. Τέσσερις μπορούν να είναι οι, εκθε... οι σελίδες της έκθεσης. Αυτοί είναι οι ισχύοντες περιορισμοί σε χαρακτήρες. Εντάξει, να μην μείνουμε και σε 4 ή 5 σελίδες, αλλά έστω 10-15 το πολύ, για να δώσουμε 4-5 βασικά πολιτικά μηνύματα σε τομείς που είναι σημαντικοί και έχουν σημασία για τους ε, συμπολίτες μας. Δεν λέω ότι υπάρχουν θέματα που δεν θα πρέπει να συμπεριλάβουμε, αλλά επειδή κάνουμε τόσα πολλά πράγματα σε τόσους πολλούς ειδικού τομείς, ε, ας προσπαθήσουμε, έλεος δηλαδή, να εστιάσουμε για τις χρονιές 15 και 16 σε λίγα και καλά. Αυτό είναι η επιθυμία μου. Ευχαριστώ. Thank you very much, Frank. I see you ended on the... Σας ευχαριστώ. Καταλήξατε στην ετήσια έκκληση για λιγότερες τροπολογίες. Να δούμε αν φέτος ε, θα λειτουργήσει. Έχουμε να κάνουμε με πολύ σημαντικά θέματα. Βεβαίω προσπαθούμε να τα ευθυγραμμίσουμε. Σας ευχαριστώ που μας αναφέρατε τα πιο ε, σημαντικά στοιχεία. Θέλει κάποιο συνάδελφο να πάρει το λόγο, κύριος Γιούρικ. Χωρίς μικρόφωνο ο μιλητής. Επαναρχόμαστε στο θέμα των θεμελιωδών δικαιωμάτων, γιατί πριν από λίγο καιρό είχαμε και την επίσκεψη του Διευθυντή ο Φλάχαρτη της, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα. Δεν θέλω να επαναλάβω τα επιχειρήματα που σας παρουσίασα στη διάρκεια εκείνης της συνεδρίασης, αλλά θα ήθελα να ευχηθώ καλή επιτυχία στην ε, κυρία Κίνγκα, γιατί θα είναι μια δοκιμή, μια δοκιμασία για τη... Ε, ε, ε τι συμβαίνει εδώ σε, αυτήν την, ε, <clears throat> σε αυτό το κοινοβούλιο. Δεν ε, θα επανέλθω σε αυτά που είπα και στον κύριο Φλάχερτη. Απλά να θυμίσω ότι επέμεινα για τη σημασία το άρθρο 2, ε, το άρθρο 2 για το δικαίωμα στη ζωή, του άρθρου 11 ε, για το άρθρο για την ελευθερία λόγου που στο θεμελιο... στα θεμελιώδη δικαιώματα αναφέρεται πολύ σωστά άμεση ελευθερία λόγου με το δικαίωμα ενημέρωσης χωρίς κανένα εμπόδιο από τις δημόσιες αρχές. Για παράδειγμα σήμερα για το θέμα της μετανάστευσης ε, στην ε, Σουηδία είδαμε ότι υπάρχει μπλοκάρισμα από πλευρά των δημοσίων αρχών εφόσον πρόκειται για ενημέρωση για ε, κλιματικές ποινικές περιοχές που συνδέονται με, ένα φαινόμενο, με το φαινόμενο της νόμιμης μετανάστευσης. Το θέμα της ελευθερίας λόγου. Άρθρο 11 συνδέεται άμεσα με το δικαίωμα στην ενημέρωση. Είναι Πτυχέ πραγματικά θεμελιώδεις. Δυστυχώ δεν έλαβα καμιά απάντηση από τον κύριο Φλάχερτη. Φλάερτη. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να αναφέρουμε αυτά τα ε, θέματα στην έκθεση που ετοιμάζουμε τώρα. Υπάρχουν και άλλες πτυχέ, όπως ας πούμε το δικαίωμα στην παιδεία στο άρθρο 14 που επίσης δέχονται επιθέσεις και που τα εγγυώνται τα κράτη, αλλά συχνά παραβιάζονται. Υπάρχουν πραγματικά προβλήματα λοιπόν εφόσον πρόκειται για θεμελιώδη δικαιώματα. Ίσως να μην συμφωνούμε εάν πρόκειται για μια χώρα όπου κινδυνεύουν αυτά τα δικαιώματα, αλλά σίγουρα συμφωνούμε ε, εφόσον πρόκειται για παραδείγματα. Γιατί το πρόβλημα υπάρχει και είναι πολύ σοβαρό. Και αν υπάρχουν προβλήματα που διαπιστώνονται παντού, θα πρέπει να το συζητήσουμε. Κατά τη γνώμη μου, αυτή η έκθεση θα είναι μια μεγάλη δοκιμή για το αν υπάρχει δυνατότητα ανοιχτού διαλόγου, ανοιχτή συζήτηση και ε, ειλικρινού συζήτηση στο κοινοβούλιο μας γύρω από τα θέματα που πραγματικά, όχι μόνο όνομα, είναι πραγματικά ουσιαστικά και θεμελιώδη. Καταρχά πρέπει να ευχαριστήσουμε τον εισηγητή και τους κοιόδες για αυτήν την παρουσίαση και το σχέδιο για την έκθεση για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Εγώ από ό,τι κατάλαβα η έκθεση αυτή θα αποτελέσει μια νέα προσέγγιση σε σύγκριση με παλαιότερες εκθέσεις. Και νομίζω πως είναι καλή ιδέα να προσπαθήσουμε να εστιάσουμε στα πιο σημαντικά θέματα. Και κράτος δικαίου είναι θεμελιώδες σημασία όχι μόνο για την Ουγγαρία και την Πολωνία, αλλά γενικώ παντού Είπατε ότι θα χρειάζεται να γίνει ένας μακρύς κατάλογος ομάδων και φαινομένων και τέτοια. Αλλά είναι σημαντικό να μάθουμε τη σημασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των διαφόρων δικαιωμάτων των μειονοτικών ομάδων. Δεν είναι απαραίτητο να μιλήσουμε για τους Ρωμά, τους Εβραίους ή τους LGBT, αλλά εν πάση περιπτώσει να πούμε ξεκάθαρα ότι κάθε μειονότητα πολιτιστική, ε, θρησκευτική, ε, εθνοτική έχουν το ίδιο δικαιώματα Είμαι βέβαιο ότι ο, έκθεση, εισηγητής και οι σκιώδες θα λάβουν υπόψη αυτή την προσέγγιση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πίτερ. Η Σεσίλ Έγκαι. Σας ευχαριστώ, Κλόντο. Πρέπει να πω ότι, ότι με σλίβει. Μάλλον χαίρομαι για τη διαφορετική δομή που πρότεινε ο εισηγητής και τον ευχαριστώ για αυτή την προσπάθεια. Σημερίζομαι την προοπτική για το γεγονός ότι το ψήφισμα του Κοινοβουλίου να μην μείνει ε, ένα απλό ψήφισμα που δίνει πληροφορίες. Πρέπει να προσπαθήσουμε να το ξεπεράσουμε αυτό. Αυτό το κείμενο θα πρέπει να ενσωματωθεί χωρίς να επικαλύπτει άλλες εκθέσεις που ασχολούνται με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ωστόσο, η σύνθεση δεν πρέπει να γίνει εις βάρος ε, του περιεχομένου και της ορθότητας των ε, πληροφοριών. Καλό λοιπόν τον εισηγητή σε αυτό το σημαντικό ε, σημείο να, να μην, να μην επιβαρύνουμε το περιεχόμενο και τις πληροφορίες. Όντως θα πρέπει κάποια στοιχεία να, ε, να δυναμωθούν. Τα κύρια στοιχεία αφορούν τις παραγράφους που αναφέρονται στην ε, μετανάστευση. Διάβασα με πολύ προσοχή και πιστεύω πως η ορολογία που χρησιμοποιεί ο εισηγητής δεν είναι πολύ σαφής. Δεν λαμβάνει επαρκώς υπόψη τη θέση του Κοινοβουλίου, κυρίως για ορισμένα προϋπάρχοντα ψηφίσματα όπου εστιάζεται αποκλειστικώς στην Αφρική και νομίζω πως αυτό δεν είναι σωστό. Και εδώ θυμίζω μιλάμε για τα θεμελιώδη δικαιώματα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, επί τη ουσία των τροπολογιών που θα υποβάλω ε, στο όνομα της ε, ομάδα μου είναι το πρώτο σημείο αυτό τη μετανάστευση. Ένα σημαντικό στοιχείο, τροποποίηση τη παραγράφου 8 του σχεδίου έκθεση όπου η συγκητή συζητά συγκεκριμένη διάκριση ανάμεσα σε οικονομικούς μετανάστες και πρόσφυγε. Θέλω να επιμείνω για το γεγονό ότι όσον αφορά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αυτή η διάκριση είναι εκτό θέματο Γιατί, Γιατί εδώ πρόκειται για την έκθεση για τα ανθρώπινα ανθρώπινα δικαιώματα και θα ήθελα να δω κάτι το οποίο να ε, τα ξεπερνά αυτά. Πριν από λίγα λεπτά και πριν από λίγες ώρες ακούσαμε την έκθεση για το Global Compact και για το, τις δηλώσεις της Νέας Υόρκης. Ένα έγγραφο το οποίο προβλέπει προστασία όλων των μεταναστών ανεξάρτητα από το νομικό τους καθεστώς. Αυτό ε, λέγεται και στα έγγραφα που έχουμε και θα μπορούσαμε έτσι να κάνουμε ένα άλμα ακόμα, να είμαστε πιο φιλόδοξοι. να μιλάμε ε, ας πούμε κυρίως για τα δικαιώματα όχι μόνο στα, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης αλλά και, και επιγραμμικά και ε, στα υπόλοιπα μέσα ε, να θυμίσω και για τα fake news αλλά και για το θέμα των διακρίσεων νομίζω πως είναι απαραίτητο να ενταχθούν συγκεκριμένες παραπομπές σε σχέση με ειδικέ μορφές διακρίσεων που δεν αναφέρονται ρητά. Και εδώ πιστεύω πως στη συζήτηση εδώ αναφέρθηκαν, δηλαδή αντισημιτισμός, ισλαμοφοβία, αντιαθηγανισμός και τα λοιπά. Ε, κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντός της Ένωσης είναι κρίσιμη, πρέπει να είμαστε άγρυπνοι και να καταγγέλουμε τις παραβιάσεις και να προτείνουμε καινοτόμε λύσεις. Κλείνω γιατί αυτά είναι μόνο κάποια, κάποιες από τις τροπολογίες που θα υποβάλω. Υπάρχουν όμως και ένα σωρό άλλα σημεία και θα προσπαθήσω στο μέτρο του δυνατού να ε, ακολουθήσω τη θέση του εισηγητή, τη στάση μάλλον του εισηγητή. Ευχαριστώ, Σεσίλ. Να κλείσουμε εδώ, διότι δεν έχουμε πολύ χρόνο. Πάντα σκέφτομαι ότι αυτή είναι μια από τις δύσκολες εκθέσεις. Αρχικά φαίνεται πάντα ελκυστικά εύκολη, αλλά δεν είναι. Πάντα είναι δύσκολη, διότι όπως βλέπετε ήδη από τη συζήτηση αυτή, θα πρέπει να εξεταστούν όλες οι παράμετροι και όπως ε, περιέγραψε και ο εισηγητής και οι συνάδελφοι φαίνεται πως είναι δύσκολο το θέμα. Λοιπόν, 27 Οκτωβρίου είναι η προθεσμία κατάθεσης ε, τροπολογιών. Ο εισηγητή περιέγραψε τις βασικές παραμέτρους, αλλά αυτό ποτέ δεν ε, εμποδίζει κανέναν να υποβάλει τροπολογίες. Ε, πειθαρχία απαιτείται λοιπόν. Να προσπαθήσετε να παρουσιάσετε με απλό τρόπο αυτά που θέλετε και να επικεντρωθείτε στα απαραίτητα. Και κατόπιν να εξετάσουμε τις ε, διάφορες άλλες σχετικές εκθέσεις. Νομίζω πάντως ότι το θέμα βρίσκεται σε καλά χέρια, ε, στα χέρια του κυρίου Έγκελ. Φρανκ, ε, θέλεις να πεις τίποτα άλλο πρώτο να προχωρήσουμε. Πολύ σύντομα, Κλόντα, μου επιτρέπεις, ευχαριστώ και πάλι για αυτόν τον γύρο συζήτησης. Ε, φυσικά γνωρίζω πολύ καλά ότι θα υπάρξουν προσπάθειες να παρουσιαστεί με πιο απλό τρόπο το θέμα αυτό. Όλα εξαρτώνται από ε, το πόση όρεξη έχουν οι άλλοι να επαναφέρουν όλα τα θέματα ή όχι. Ε, βέβαια γνωρίζω πολύ καλά ότι κάθε συνάδελφος έχει το δικαίωμα να υποβάλει όσες τροπολογίες θέλει. Εγώ ελπίζω να μην καταλήξουμε με χίλιες τροπολογίες όπως έχουμε δει στο παρελθόν. Και να έχουμε ε, σχεδόν τηλεφωνικό κατάλογο στις, ε, στην Ολομέλεια. Στον ε, συνάδελφο Γιούρεκ να πω ότι δεν έχω αντίρρηση σε μία συζήτηση για όλα τα θέματα, αλλά θα πρέπει αυτό να γίνει στο σωστό πλαίσιο. Δεν μπορούμε να αγνοούμε το κράτος σε δικαίου και να κρυβόμαστε πίσω από τρία-τέσσερα άρθρα τριών-τεσσάρων ε, ε, επισήμων ε, εγγράφων. Γνωρίζω πολύ καλά τι είναι το δικαίωμα στη ζωή. Ξέρω όμως ότι αυτό δεν μπορεί να αποτελεί λόγο για ρελατιβισμό, να περιορίζουμε το δικαίωμα λόγου οποιοδήποτε. Πάντως σίγουρα μπορούμε να τα συζητήσουμε όλα. Επίσης να πω ότι όσον αφορά τις μειονότητες. Γνωρίζω ότι δεν έχω θίξει καθόλου το θέμα αυτό στο σχέδιο της έκθεσης. Ε, καταλαβαίνω ότι θα πρέπει να ενσωματωθεί. Περιμένω λοιπόν να δω τις τροπολογίες, μπορώ να υποβάλω κι εγώ κάποιες. Και ξέρω ότι και άλλοι συνάδελφοι θα επικεντρωθούν στο θέμα αυτό. Πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να βρούμε ε, τρόπους ε, διατύπωσης ε, για να τα περιγράψουμε αυτά. Και στη Σεσίλ θα ήθελα να πω ότι για, κατά τη γνώμη μου προφανώς υπάρχει χώρος για συζήτηση και μπορούμε να διατυπώσουμε κάθε παράγραφο με διαφορετικό τρόπο. Εγώ δεν είμαι αντίθετο στο να τα συζητήσουμε όλα. Δεν είμαι αντίθετο σε οποιαδήποτε διαφορετική προσέγγιση και για οποιαδήποτε πτυχή. Δεν υπάρχει λοιπόν μεγάλο πρόβλημα στην αντιπαράθεση και στη σύγκριση κειμένων που θα ήθελες να υποβάλεις. Για μένα ένα πράγμα είναι σαφές ότι αν κάνουμε διάκριση ανάμεσα σε όσους έρχονται εδώ χρήζοντας βοηθείας και εκείνος που δεν χρειάζονται καμία προστασία αλλά ελπίζοντας θα βρούνε καλύτερη ζωή εγώ δεν λέω πως δεν είναι απαραίτητο να προστατευτούν και οι δύο κατηγορίες. Δεν το έχω πει, δεν το έχω γράψει και αν νομίζεις πως ε, αυτό έχω γράψει, τότε θα το διατυπώσουμε διαφορετικά, ώστε να μην βγαίνει τέτοιο νόημα. Αυτά. Έχω να πω και θα περιμένουμε τις τροπολογίες και θα τις διαχειριστούμε. Η 27 Οκτωβρίου είναι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Ωραία, πάμε στο σημείο 17 και είναι η έκθεση της Άννας Μαρία Κοράτσα Μπίλτ. Και πριν ξεκινήσουμε θα ήθελα να καλωσορίσω μια οργανώση νέων από τη Σουηδία MUF αν δεν κάνω λάθος. MUF. Δεν ήθελα να το προφέρω λάθος. Σας καλωσορίζουμε θέρμα και σας κάλεσε βεβαίως η κυρία Κοράτσα. Πείτε, είστε ευπρόσδεκτοι στην συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Και εδώ έχουμε να εξετάσουμε την έκθεση της κυρίας Κοράτσα. Πείτε και το ψήφισμα της 11 Μαρτίου σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών. Η προθεσμία για τη μεταγραφή αυτού του νομοθετήματος εξέπνευσε από το 2013 και θέλουμε να εξετάσουμε το πλαίσιο ε, εφαρμογής αυτής της οδηγίας. Η κυρία Κοράτσα Μπίλτε υπέβαλε ένα σχέδιο έκθεσης πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές και τώρα θα συζητήσουμε τις τροπολογίες. Με τα χαράς λοιπόν θα συζητήσουμε αυτές τις τροπολογίες και μετά πρώτα η συγγήτρια και μετά οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι φρικτό έγκλημα κακοποίηση παιδιών ε, μέχρι και βρεφών ε, που είναι τα πιο ευάλωτα μέλη της κοινωνίας από ε, σωματική, ψυχολογική μέχρι online είναι αυτή η βία και έχουμε την σεξουαλική κακοποίηση τέτοια εγκλήματα τα οποία διαδίδονται, παρουσιάζονται και πληρώνουν κάποιοι. Είναι ένα πάρα πολύ κερδοφόρο ε, επάγγελμα εντός και υπάρχουν και οι ε, οι χώροι όπου γίνεται chatting ε, με, με θέματα αυτά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ζήτημα. Πρέπει να πούμε ότι είναι επιτετευμένα τα μέσα τα οποία χρησιμοποιούνται. Η οδηγία που υιοθετήσαμε τη Δευτέρα, κάποιοι ήσασταν εκεί, το 2011 είχαμε πετύχει ένα ιστορικό επίτευγμα με την οδηγία Όταν μιλάμε για διασυνοριακά εγκλήματα, χρειάζεται και διασυνοριακή αντιμετώπιση. Προβλέπονται ελάχιστα ε, μέτρα κατά πολέμησης των κακοποιήσεων, ορίζεται το αδίκημα και υπάρχουν μέτρα κατά πολέμησης της ατιμορρησίας και προστασίας των παιδιών. Ε, έχουμε λάβει από την Κομισιόν δύο εκθέσεις υλοποίησης. Είχαμε τρεις ακροάσεις, Λιμπελκ και σκιώδεις ηγητές, ήρθαν εμπειρογνώμονες, διάφοροι άλλοι από την κοινωνία των πολιτών, από τις αρχές επιβολής νόμου στα κράτη-μέλη. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ τους σκιώδεις γιατί είχαμε εξαιρετική συνεργασία. Μελετήσαμε σε βάθος το θέμα. Θέλω να τους συμπεριλάβω όλους και το ίδιο θα προσπαθήσω να κάνω και με τις συμβαστικέ τροπολογίες τις οποίες και επεξεργαζόμαστε τώρα. Ποιος είναι ο στόχος της έκθεσής μας είναι να δούμε κατά πόσον τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν ε, σωστά και πλήρως την οδηγία. Ποιες είναι οι λήψεις και αυτό που θέλουμε επίσης είναι να διατυπώσουμε συστάσεις για το πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί η εφαρμογή της οδηγίας. Μιλήσατε για τις τροπολογίες, είναι 160 και πολλές από αυτές ε, είναι πιο πολύ επικριτικές προς την Κομισιόν ε, που ουσιαστικά δίνει βάρο στι εκθέσει τη στην μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και στην εφαρμογή τη οδηγία. Έχω καταθέσει κάποιε τροπολίε, αλλά θέλω να πω ότι η εστίαση ίσω θα πρέπει να είναι περισσότερο στο επίπεδο των κρατών μελών. Και όχι να κατηγορείται η Κομισιόν, γιατί η οδηγία τελικά δεν υποχρεώνει πραγματικά τα κράτη-μέλη να παρέχουν στατιστικά στοιχεία. Επομένω, ε, μία μελλοντική αναθεώρηση. Δεν το ζητώ αυτό τώρα. Μπορούμε να το δούμε και μπορεί να θελήσουμε να καταστήσουμε υποχρεωτική την ε, παροχή στατιστικών στοιχείων, αλλά στην έκθεση αυτή προ το παρόν μπορούμε να στήσουμε από τα κράτη-μέλη σίγουρα να συνεργάζονται καλύτερα και περισσότερο μεταξύ του ε, και να δίνουν και στην Κομισιόν ε, τα στατιστικά αυτά στοιχεία και προσβλέπουμε και σε μια επόμενη πληρέστερη έκθεση από πλευρά Κομισιόν. Για τι υπόλοιπε τροπολογίε, ε, κύριε Πρόεδρε, εγώ ακολουθώ την δομή τη οδηγία έτσι, γιατί μιλάμε για θέμα ποινικού δικαίου και είναι τεχνικό πολύπλοκο το θέμα για το ουσιαστικό ποινικό δίκαιο. Προτείνω ε, μια τροπολογία, όπως και πολλοί άλλοι συνάδελφοι, που τροποποιεί τον όρο της παιδικής πορνογραφίας και μιλάμε για υλικό παιδικής σεξουαλικής ε, κακοποίησης, για να μην υπάρχει διπλή θεματοποίηση. Είναι θέμα συνένεσης. Η παιδική πορνογραφία ε, είναι σαν να συνεπάγεται την συνένεση. Ζητούμε λοιπόν να αντικατασταθεί αυτός ο όρος ε, και από πολιτικές πλευράς αυτό είναι σημαντικό. Δεν σημαίνει ότι μειώνεται το πεδίο εφαρμογής όταν μιλάμε για υλικό παιδικής ε, σεξουαλικής κακοποίησης, γιατί αυτό περιλαμβάνει και αυτά που λέει η οδηγία για την ε, παιδική πορνογραφία. Λυπούμε που είμαι τεχνική, αλλά ε, σας δώσω ένα παράδειγμα. Το, το δίκτυο παιδο, παιδεραστών χρησιμοποιεί και φωτογραφίες παιδιών που μπορεί να έχουν ποστάρει γονείς τους στο διαδίκτυο ή που να τα, μπορεί να τα βρει κανείς σε ιατρικά αρχεία. Όταν χρησιμοποιούνται, γίνονται, ε, η χρήση τους δηλαδή γίνεται ποινική, αξιόπινη πράξη, ενώ δεν ήταν αρχικά. Επίσης, το επιβαρυντικά μέτρα όταν η σεξουαλικοποίηση διαπράτεται από έναν κοντινό ε, του παιδιού. Συνήθως το άτομο που υποτίθεται ότι εμπιστεύεται το παιδί, που έχει την εξουσία, που είναι αυτός που θα έπρεπε να φροντίζει το παιδί, είναι αυτός που διαπράττει και για σειρά ετών ε, τα εγκλήματα αυτά. Επίσης, δεν υπάρχει υποπτία πολλές φορές και αυτό διευκολύνει τη διαπράξη των εγκλημάτων αυτών. Νομίζω επίσης πρέπει να περιλάβουμε και για το μέλλον ε, έναν επικαιροποιημένο πίνακα τέτοιων εγκλημάτων όπως είναι ο εξαναγκασμός, ε, η τα κτλ. Ε, και ιδίως ε, στο διαδίκτυο. Βλέπουμε να αυτοκτονούν στο facebook ε, νεαρά κορίτσια γιατί δεν μπορούσαν να βγάλουν φωτογραφίες που είχαν αναρτήσει πρώην σύντροφοί τους στα, στο facebook για να τις εκδικηθούν και, και μετά σχολίαζαν οι άλλοι φίλοι και δεν μπορούσαν να το αντέξουν αυτά τα κορίτσια. Και έρχομαι στο δεύτερο σημείο της οδηγίας που είναι η έρευνα και δίωξη. Εδώ θέλω να υποστήριξω όλε τι τροπολογίε των συναδέλφων που ζητούν από τα κράτη-μέλη να αξιοποιήσει όλα τα εφιστάμενα εργαλεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχει το ένδαλμα ε, ερευνά η Europol και η Eurojust κάνουν πολύ καλή δουλειά για την καταπολέμηση των ε, εγκληματικών δικτύων. Η Europol και η Eurojust πρέπει να έχουν και του απαιτούμενου πόρου στη διάθεσή του για να μπορέσουν να φέρουν σε πέρα στην αποστολή του και να αξιοποιήσουν καλύτερα τι κοινέ ε, ομάδες έρευνας. ό,τι αφορά τη βελτίωση ανταλλαγή πληροφοριών είναι σημαντικό αυτό και η διαλειτουργικότητα των βάσεων δεδομένων κάτι που προτείνουμε. Σε ό,τι αφορά την πρόληψη πρόληψη, υπάρχουν κάποια προγράμματα πρόληψης και παρέμβασης για άτομα που ενδεχομένως στο μέλλον να διαπράξουν αδικήματα σεξουαλικά σε βάρος παιδιών ή άλλο θέμα εκπαίδευση των αξιωματούχων, των διαφόρων ε, και ευαισθητοποίηση των παιδιών. Πολύ σημαντικό για το διαδίκτυο. Και τα κράτη-μέλη θα πρέπει στην νομοθεσία τους υποχρεωτικά να συμπεριλάβουν ελέγχους του ε, παρελθόντος, του ιστορικού, ατόμων που εργάζονται σε τομείς που έχουν να κάνουν με παιδιά και που έχουν πρόσβαση στα παιδιά. Βελτίωση συλλογή δεδομένων επίσης ε, σε εθνικά ε, μητρώα για να δούμε τι ποινικέ καταδίκες υπάρχουν ε, και να εντοπίσουμε τους θύτες για να μην υπάρξει υποτροπή και διαπράττουν συνεχώ τα ίδια Υπάρχουν κάποια helplines, πάρα πολύ ε, καλή δουλειά που κάνουν αυτές οι τηλεφωνικές γραμμές βοήθειας. Άλλο θέμα είναι αποφυγή της διπλής θυματοποίησης και της ε, κατηγορίας των ίδιων των ε, θυμάτων τελικά. Άρθρο 15. Είναι λίγο επίμαχο. Έχω καταθέσει και εγώ τροπολογίες. Θα υποστηρίξω και τις τροπολογίες των συναδέλφων σε ό,τι αφορά την απομάκρυνση στην πηγή του υλικού αυτού ε, είναι προτεραιότητα. Όχι το μπλοκάρισμα, την ε, απόσυρση θέλουμε αυτού του υλικού. Το μπλοκάρισμα θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν δεν είναι δυνατή η απομάκρυνση και επίσης θα πρέπει να βελτιωθεί η συνεργασία των κρατών με τον κλάδο, με τα δίκτυα, τα κοινωνικά, με τις πλατφόρμες και με τους τρίτους, τις τρίτες χώρες ε, όταν η πλατφόρμα βρίσκεται εκτός ένωση, Θα πρέπει να επικαιροποιούνται οι μαύρες λίστες που έχουμε σε επίπεδο επεξένωσης για παιδική πορνογραφία και να υπάρχει ανταλλαγή των στοιχείων με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταπολέμησης του Κυβερνογκλήματος, τη Europol και τα κράτη-μέλη. Επίσης έχουμε συμπεριλάβει κάποιες διατάξεις ώστε οι πάροχοι υπηρεσιών στο διαδίκτυο θα πρέπει να αναφέρουν στις αρχές επιβολής του νόμου το υλικό ε, παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης ε, που έχουν ε, εντοπίσει. Γιατί πράγματι είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνεται αυτό επί εξωτράωρου βάσεως. Το θέμα είναι όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να μπορεί να απομακρύνεται αυτό το υλικό και τα hotlines να έχουν το, τους απαραίτητους πόρους. Ολοκληρώντας, θέλω οπότε πάρα πολύ σημαντικό να εφαρμόσουν τα κρατημέλη την οδηγία με όλα τα μέσα που έχουν στη θέση τους και προβλέποντας κάπως, προκαταλαμβάνοντας και τις μελλοντικές εξελίξεις. Και ιδίως στον τομέα της τεχνολογίας. <laughs> Αν μπορούν οι εγκληματίες να κάνουν κάτι, πρέπει και εμείς να μπορούμε να το κάνουμε. Άρα να έχουμε τα πιο καινοτόμα μέσα για τον εντοπισμό των ε, εγκληματιών στο διαδίκτυο. Περιμένω τώρα να ακούσω τους κοιότες και βέβαια να συνεργαστώ μαζί τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Άννα Μαρία. Κατερίνα, θα μιλήσεις εκ μέρους ε, του S&D ως και συγγετρία. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα πάρω εγώ τον λόγο για να ευχαριστήσω τη συνάδελφο. Κοράτσα Μπίλτ και όλους τους κοιόδης ε, που εργάστηκαν για αυτή την έκθεση γιατί πρόκειται για ένα θέμα που πρέπει οπωσδήποτε να το εξετάσουμε λόγω του ότι είναι τόσο λεπτό και γιατί είναι σημαντικό να προσφέρουμε σε όλες ε, τις, τα παιδιά την ε, ε, την προστασία από τέτοιου κινδύνους, αλλά και να ενημερώσουμε για τους κινδύνους που προέρχονται από ε, το δίκτυο. Να ευχαριστήσω λοιπόν την κυρία ε, Κοράτσα Μπίλτε και για την προσπάθεια που έκανε για να παρουσιάσει τις πολλές και διάφορες τροπολογίες που έλαβε. Εγώ θα σταθώ σε κάποια σημεία. Εκτίμησα πολύ και στήριξα την τροπολογία που ε, υποβλήθηκε για να αλλάξει ο όρος παιδική πορνογραφία και να μετατραπεί σε μια μια άλλη και πιο κυριολεκτική φράση ε, που είναι υλικό που ε, σχετίζεται με την, παιδική, με την εκβεσική εκμετάλλευση και την παιδική πορνογραφία. Ακριβώς για να μην υπάρξει καμία ε, τέτοια προκατάληψη και ζημιά. Και αυτό διέπει και την βασική εργασία που έκαναν οι συνάδελφοι. Πρέπει να υπάρξει μια πολιτιστική αλλαγή, αλλαγή νοοτροπίας, διάχυτη, για να αποφευθεί κάθε είδους κάθε είδος ε, κατηγορία ας πούμε εναντίον των παιδιών που έχουν πέσει θύματα τέτοιων ε, αδικημάτων ε, θυματοποίηση δηλαδή δευτερογενής γιατί είναι ήδη αρκετά μεγάλα τα τραύματα που, στα οποία υπόκειται τα παιδιά Κάτι ακόμα, το οποίο συνδέεται και αυτό με την ιδέα της ε, πολιτιστικής αλλαγής, είναι και ανάγκη που υπογραμμίζεται ε, μέσα από τις τροπολογίες, ανάγκη να φτιαχτούν προγράμματα εκπαιδευτικά πρόληψης, να παρα... όντως να δοθούν στα παιδιά όλες οι δυνατότητες προστασίας, αλλά και μέσα από αυτές να υπάρξουν και τα μέσα, να, να έχουν τα παιδιά τα μέσα για να αποφύγουν αυτούς τους κινδύνους, δηλαδή να γνωρίζουν πώς να χρησιμοποιήσουν το δίκτυο με υπεύθυνο τρόπο, γιατί αυτό είναι το πρώτο μέσο για να προστατευθούν, πέρα βέβαια από το ίδιο είδος παιδείας και εκπαίδευσης που θα πρέπει να στραφεί προς τους ε, γονείς ή τους κηδεμόνες ώστε να μπορούν να προστατεύσουν και αυτοί με τη σειρά τους τα παιδιά τους από τους κινδύνους του διαδικτύου. Κάλλη μια πτυχή που θέλω να τονίσω γιατί είναι πολύ σημαντική, είναι αυτή που σχετίζεται με την ανάγκη στήριξης των κρατών, της κατεύθυνσης των κρατών προς μια πλήρη συνεργασία, γιατί ε, δυστυχώς πολλές φορές τέτοια δίκτυα περνούν από τα δίκτυα και είναι και διασυνοριακά. Η συνεργασία εδώ είναι λοιπόν απαραίτητη, όπως είναι απαραίτητο να κατευθυνθούν τα κράτη και να έχουν και τους πόρους ε, για να εξοπλιστούν ώστε να μπορέσουν να έχουν τα απαραίτητα μέσα πληροφορικής για να μπορούν να συλλέξουν ηλεκτρονικές αποδείξεις γιατί αυτού του είδους τα δικήματα γίνονται μέσα από το δίκτυο και άρα λοιπόν τα κράτη πρέπει να έχουν στη διαθεσή τους τις καινοτόμες λύσεις για να μπορέσουν ακριβώς να διώξουν τέτοιου είδους ε, αδικήματα και τους υπευθύνους online. Τέλος, αυτό που είναι επίσης σημαντικό και εδώ έχει σκόπο μα συμπεριληφθεί είναι η στήριξη στα παιδιά θύματα τέτοιων μεγάλων αδικημάτων και σοβαρών αδικημάτων. Ευχαριστώ του συναδέλφου και εκφράζω την πλήρη μου στήριξη στην εργασία που έχει γίνει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ Κατερίνα, ο κύριος Γιούρεκ. Ευχαριστώ πολύ. η σεξουαλική κατομεταχείριση παιδιών ε, και η διάδοση οποιασδήποτε τέτοιας ε, συμπεριφοράς ε, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να καταπολεμήσουμε. Ευχαριστώ πολύ την Άννα Μαρία Κορατσαπίλτ για το θέμα αυτό, διότι έχουμε να κάνουμε με ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα, διασυνοριακή εγκληματικότητα και το διαδίκτυο, όπως όλοι γνωρίζουμε, δεν έχει σύνορα. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να εμβαθύνουμε στο θέμα. Οι τροπολογίες μου θέτουν το θέμα αυτό σε ευρύτερο πολιτιστικό πλαίσιο. Έχουμε τη σύμβαση της Γενέβης που υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να καταπολεμούν την πορνογραφία, την παιδική πορνογραφία. Αλλά τα κράτη δεν συμμορφώνονται με αυτές. Επίσης, Όσον αφορά τις διατάξεις για τη διασυνοργική τηλεόραση, επίσης ε, υποχρεώνει ε, να καταπολεμηθεί η ε, παιδική πορνογραφία, αλλά ούτε με αυτές τις διατάξεις σε συμμορφώνονται όλοι. Ο Γιώσεφ Φρίτσλα από την Αυστρία ήταν ήταν ε, ε, ε, παιδόφιλος και σε παθολογικό βαθμό έβλεπε παιδική πονογραφία και κατόπιν τα έκανε και μόνος του. Πρέπει λοιπόν να ξεφύγουμε από αυτήν την μαζική κουλτούρα παιδικής πορνογραφίας που παραβιάζει κάθε αίσθηση αξιοπρέπειας. Αυτό λοιπόν διότι η παιδική πορνογραφία οδηγεί σε αυτό που είπε η Άννα Μαρία Κορατσαπίλτ, ε, καλούνται κορίτσια να κάνουν κάτι στο πλαίσιο μιας σχέσης ε, και κατόπιν ε, αυτά δημοσιεύονται. Πρέπει λοιπόν να εξαλείψουμε τις αιτίε των πράξεων αυτών. Ευχαριστώ πολύ. Άννα Μαρία, να σου ξαναδώσω το λόγο για να συνοψίσεις, σε παρακαλώ. Ψηφοφορία στην Επιτροπή στις 21 Νοεμβρίου, στις 13 Νοεμβρίου, συγγνώμη. Θέλεις και εσύ να παρέμβεις, ε, δεν ζήτησε το λόγο. Ήρθες ειδικά γι' αυτό, μάλιστα, παρακαλώ. Τζιν, σου δίνω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ε, είμαι βέβαιη ότι έχω πολλά να προσθέσω σε αυτά που ήδη υπόθηκαν. Νομίζω ότι η αρχική έκθεση από μόνη της ε, ήταν ένα ε, πολύ δυνατό κείμενο. Οι τροπολογίες που έχουμε υποβάλει κυρίως ε, σχετίζονται με τα δεδομένα που πιστεύουμε θα πρέπει να διατίθονται και που δεν διατίθενται. Επίσης έχουν να κάνουν με την έλλειψη συνεργασίας που φαίνεται να υπάρχει μεταξύ των κρατών μελών στον συγκεκριμένο αυτόν τομέα. Και ένα από τα θέματα που θέλαμε να θίξουμε είναι κατά την ανταλλαγή πληροφοριών ε, και μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου θέλουμε να ε, διασφαλίσουμε την ασφάλεια, την επισκεφτικότητα των ε, πληροφοριών αυτών για να μην πέφτουν σε λάθος χέρια. Επίσης, όσον αφορά το θέμα αυτό και την κακοποίηση των παιδιών, Το θέμα δεν είναι αν νιώθουμε ότι πρόκειται για πορνογραφία, το θέμα είναι να υπάρχει εφαρμογή των διατάξεων. Καταφέρνουμε να ε, περάσουμε τις ιδέες μας σχετικά με ε, ελέγχους ε, των διαφόρων ανθρώπων ε, και περιπτώσεις κακομεταχείρισης παιδιών. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό που έχουμε εδώ αποτελεί πολύ ισχυρή ανταπόκριση στην ε, έκθεση εφαρμογής ή μάλλον την έκθεση για την ε, έλλειψη εφαρμογής, διότι όλοι συμφωνούμε ότι αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό θέμα και γι' αυτό θα θέλαμε κάποια κράτη-μέλη να δίνουν τις προσπάθειές τους για να καταπολεμήσουν το φαινόμενο αυτό ε, όπως πρέπει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Τζιν. Συγγνώμη που δεν σε είδα ξανακοιτώ για να βεβαιωθώ ότι δεν υπάρχει κάποιος άλλος και που θέλει να πάρει το λόγο. Ε, εντάξει, Ανά Μαρία, θα ήθελες να συνοψίσεις. Ευχαριστώ, Κλόντ, ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Είμαι πολύ ικανοποιημένη που καταφέραμε να φτάσουμε σε ευρεία συνένεση με όλες τις πολιτικές ομάδες. Ευχαριστώ όλους τους σκιώδους, σκιώδεις εισηγητές. Ευχαριστώ και σένα, Κατερίνα όσον αφορά το θέμα της κουλτούρας, το να ενδυναμώσουμε τα παιδιά τα ίδια είναι μακροπρόθεσμα ένα πολύ ισχυρό εργαλείο για την καταπολέμηση της ε, σεξουαλικής κατοικοποίησης. Το πρόβλημα είναι στο διαδίκτυο, δεν βλέπει κανείς ε, ποιο κρύβεται από πίσω. Έχουμε λοιπόν το φαινόμενο της άγρας, ε, το οποίο δυσκολεύει πολύ, τα... δυσκολεύει πολύ την κατάσταση και συμφωνώ απολύτως ε, όσον αφορά την ε, ασφάλεια των στοιχείων. Με την έκθεση αυτή έχουμε την ευκαιρία να ασκήσουμε πίεση στα κράτη-μέλη, να τονίσουμε το πόσο επίγον είναι το θέμα και να τα καλέσουμε να ε, εφαρμόσουν πλήρως την οδηγία. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να εφαρμόσουμε την πολιτική για την καταπολέμηση της ε, σεξουαλικής κακοποίησης ε, των παιδιών στην Ευρώπη. Κάτι ακόμα, είμαι υπέρ της προστασίας του ιδιωτικού βίου και όταν ε, μιλάμε με τις αρχές επιβολής του νόμου μας μιλάνε για τις δυσκολίες στο να προστατεύσουν τα παιδιά στο διαδίκτυο διότι είναι πολύ περιορισμένα τα εργαλεία τους ενώ οι εγκληματίες χρησιμοποιούν τα πιο καινοτόμα τεχνολογικά μέσα. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε και εμείς το ίδιο. Η, η προστασία του ιδιωτικού βίου δηλαδή δεν μπορεί να μας εμποδίζει να χρησιμοποιήσουμε τεχνολογίες, να επενδύσουμε σε νέα εργαλεία για να μπορέσουμε να εντοπίσουμε στο διαδίκτυο τους εγκληματίες. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και όλους τους κοιόδης συζητητές. Σε ευχαριστώ, σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία με την έκθεση αυτή. Ευχαριστώ και τους ε, συναδέλφους και τους συζητητές. Συνάδελφοι, προχωράμε τώρα στο σημείο 19, καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου. Η συγητής είναι ο κύριος Κοράο, είναι παρόν. Έχουμε λοιπόν παρουσίαση των τροπολογιών ε, πάνω στην ε, προτινόμενη οδηγία για την καταπολέμηση της νομοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Ε, στις 28 ε, Σεπτεμβρίου ο εισηγητή παρουσίασε το σχέδιο Έκθεση. Ε, το Συμβούλιο υιοθέτησε τη γενική του προσέγγιση τον Ιούνιο του 2017. Θα θυμάστε ότι η προτινόμενη οδηγία εναρμονίζει ε, το έγκλημα της νομοποίησης παρανομών εσόδων συμπεριλαμβανομένου του θέματος των κυρώσεων και συνολικά είχαμε 182 τροπολογίες οι οποίες υποβλήθηκαν είχαν να κάνουν και με το θέμα της ε, ε, νομοποίησης ε, των ιδίων εσόδων από εγκληματικέ δραστηριότητες, τα θέματα απόδειξης, δέσμευσης και κατάσχεσης. Σε συνάδελφοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που βρίσκεστε εδώ για να συζητήσουμε το θέμα αυτό πέμπτη απόγευμα μετά από ένα πολύ γεμάτο πρωί. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την παρουσίαση εδώ και δίνω το λόγο στον εισηγητή μας, τον κύριο Κόραο. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Grazie, Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις εισηγητές για τις ε, πολυάριθμες ε, τροπολογίες που υπέβαλαν. Το περιεχόμενο ε, είναι ωστόσο πολύ τεχνικό και περίπλοκο. Λάβαμε 182 τροπολογίες, επί τη βάση των οποίων σκοπεύουμε να κάνουμε καλές συμβιβαστικές τροπολογίες. Πολλές από αυτές είναι σύμφωνες με τις θέσεις που έχουμε στηρίξει μέχρι τώρα και μάλιστα την συμπληρώνουν είναι πρόθεσή μου να ε, μαζί με τους Κιώδης ε, να βρούμε μία κοινή θέση στις συμβιβαστικέ όσο γίνεται πιο σύντομα όπως άλλωστε κάναμε και μέχρι τώρα ε, παρά τις καθυστερήσεις που είχαμε πριν από την ανάθεση αυτής της έκθεσης και το συζητήσαμε και στις προηγούμενες μας επαφές. Είμαι βέβαιος ότι θα το καταφέρουμε γιατί οι θέσεις είναι κοινέ. Οι θέσει μα είναι κοινέ. Ε, θα περιοριστώ στο να σχολιάσω κάποιε από τι τροπολογίε ανά θέμα πριν να δώσω το λόγο και στους ε, σκιώδει για αυτά που θεωρώ πως είναι τα πιο σημαντικά σημεία που θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνονται στην τελική έκθεση. Για παράδειγμα, ε, είμαστε υπέρ της συμπερίληψης των φορολογικών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 ε, αδικημάτων. Αυτά είναι αδικήματα που αφορούν την εφορία αλλά ξαναμπαίνουν στην πραγματική οικονομία με αποτέλεσμα να στρεβλώσουν τον ανταγωνισμό. Θα έχουν ένα δηλαδή πλεονέκτημα για όποιον ε, φοροδιαφεύγει και είναι εις βάρος των όσων καταβάλουν τους φόρους τους και άρα λοιπόν και αυτό το είδος αδικήματος θα πρέπει να ε, τιμωρηθεί. Για το θέμα της ανακύκλωσης εδώ θα πρέπει να μιλήσουμε για ε, έγκλημα για την ίδια την κατοχή, ας πούμε μπορεί αυτό να οδηγήσει σε τρελές καταστάσεις, μπορεί ας πούμε να ένας κλέφτης ε, που έχει κλέψει ένα ε, ποδήλατο να κατηγορηθεί για ανακύκλωση επειδή χρησιμοποιεί αυτό το ποδήλατο για να κλέψει κάποιον άλλον μετά. Εν γέννη υπάρχει συνένεση ανάμεσα στους σκιώδεις εισηγητές σε σχέση με την προσέγγιση που επιλέξαμε αρχικά. Ε, εγώ θα θέλω να διατηρήσω αυτή την προσέγγιση και στις συμβιβαστικές, δηλαδή η ιδέα μας να παραμείνει δηλαδή ένα είδος μιας διπλής ε, οδού για να εγγυηθούμε τα δικαιώματα αλλά και να μπορέσουμε να τιμωρήσουμε την ανακύκλωση από πολύ σοβαρά δικήματα όπως το εμπόριο ανθρώπων, εμπόριο ναρκωτικών κτλ. Σε ορισμένες περιπτώσεις θα αρκεί να περιλαμβάνεται αυτό το συγκεκριμένο αδίκημα ως αδίκημα ε, όπως και η ανακύκλωση. Όσον αφορά τις κυρώσεις διαπιστώνω με χαρά ότι οι τροπολογίες των σκιωδών έχουν, ε, έχουν στόχο να αυξήσουν τη μέγιστη ποινή αλλά και τη ε, μίνιμουμ ποινή αλλά και να μιλήσουμε και για τις επιβαρυντικές περιστάσεις αλλά και να μιλήσουμε και για πρόσθετες ποινές που έχουν προταθεί όπως ας πούμε απαγόρευση από δημόσιες θέσεις ή απαγόρευση ε, να αναλάβει κανείς δημόσιες θέσεις ή ε, να ε, είναι υποψήφιος σε εκλογές. Θα πρέπει ε, επίση να υπάρχουν οι κατάλληλοι πόροι, να προβλεφθούν οι κατάλληλοι πόροι, ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν οι νέε ε, προσ... Ε, προκλήσει όπω η κυβερνοεγκληματικότητα ή η χρήση εικονικών νομισμάτων. Η συζήτηση για τι συμβιβαστικέ θα περιλάβει και τη συζήτηση για το, τη συζήτηση για το κατά πόσο το αδίκημα της ανακύκλωσης θα θεωρηθεί δόλος ή όπως εμείς θέλουμε ή αν θα θεωρηθεί και σοβαρό αδίκημα όπως προτείνει κάτι ποιος άλλος. Ε, κατά τη γνώμη μας θα πρέπει να μείνει μόνο ε, ως ε, δόλος γιατί διαφορετικά μπορεί να ανοίξει πολύ η ερμηνεία. Βέβαια, ε, είμαστε ανοιχτοί σε μια συζήτηση που θα γίνει τελείως νομικής φύσης βέβαια όσον αφορά το ορισμό, το, το πιο μέχρι που είναι η ε, ενοχή και από που και πέρα ε, αρχίζει και ο δόλος. Τώρα, στο τελικό κείμενο, τα διαδικαστικά δικαιώματα ε, ε κατηγορίας των, ε, των καταδικασμένων θα πρέπει πάντοτε να μπορεί να συζητηθεί όταν, ας πούμε, έχουν κοινωνική συμπεριφορά που είναι αυλαβής ή η αγορά αγαθών και υπηρεσιών για την ικανοποίηση πρωταρχικών αναγκών ε, ή αγορά υπηρεσιών και αγαθών που έχει δικαίωμα δικαίωμα το άτομο να αγοράσει. Ευχαριστώ και πάλι όλους όσους υπέβαλαν τροπολογίες. Εύχομαι ότι θα μπορέσουμε σύντομα να φτάσουμε σε συμβιβαστικές. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κορά και θα ακούσουμε και τους κοιόδες εισηγητές. Από το ΕΛΚ, η κυρία Χολμάιερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω θερμά του συναδέλφους, ε, βέβαια και τον εισηγητή πρώτα απ' όλα, αλλά ενώ και τους ε, σκιώδεις, ε, όπως επίσης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πολύ καλή εντατική συνεργασία. Διάβασα τις τροπολογίες συνολικά και πραγματικά νομίζω ότι ευτυχώς για το μεγαλύτερο μέρος τους ε, υπάρχει συνένεση. Υπάρχουν κάποιες αποχρώσεις ε, που εμείς έχουμε κάποια αιτήματα επιπρόσθετα, αλλά οι περισσότερες τροπολογίες είναι πολύ λογικές. Ό,τι αφορά τη συνένεση να έχουμε αυτή την ε, ε, ελάχιστη ποινή και να υπάρχει αυτή η δυνατότητα να δούμε κατά πόσο ε, θα είναι πρόστιμο αυτή η ποινή ή αν θα είναι φυλάκιση ε, γιατί σε κάποιες περιπτώσεις θα πρέπει να μην καλύπτεται μία ποινή από ένα πρόστιμο απλά αλλά να υπάρχει και μία ελάχιστη ποινή. Έχουμε επίσης την οδηγία του 2014 για την κατάσχεση, τη δίμευση ε, στοιχείων που προέρχονται από παράνομη δραστηριότητα. Νομίζω ότι είναι θετικά όλα αυτά. Σε πολύ μεγάλο βαθμό πιστεύω έχουμε καταφέρει να καταλήξουμε σε λογικές λύσεις. Έχω κάποια φυλακτικότητα και είναι κάπως διαφορετική προσέγγιση μου στο εξής όμως θέμα, κατά πόσον ε, είναι σωστή η, η προσέγγισή σας για την... το βάρος απόδειξης. Ας πούμε ότι βρίσκει στο λογαριασμό του χρήματα κάποιος και πρέπει να δικαιολογήσει από πού τα βρήκε. Ναι, εντάξει, όμως σε κάποιες περιπτώσεις ε, μπορεί να μην φέρει το όνομά του, να μην είναι ο δικαιούχος ε, ή να είναι και σε ένα άλλο κράτος ε, δικαιούχος και δεν μπορεί να αποδείξει αυτό το άτομο ότι δεν είναι δικός του ο λογαριασμός. Ξέρω και από την οικογένειά μου και στη Γερμανία ε, είχαμε 12 χρόνια έναν, αδρανή, ε, ανενεργό λογαριασμό και μάλιστα και στο Λίχνεστάιν και στον Καναδά και στην Ελβετία προσπαθούμε να ε, μπορούν να επιβεβαιώσουν οι τράπεζες να πιστοποιήσουν ότι δεν ανήκει στον τάδε ο λογαριασμός και το θέμα είναι ότι δεν το ξέρουν κάποιοι. Δεν είναι ότι δεν θέλουν να δώσουν το πιστοποιητικό, απλά δεν γνωρίζουν ούτε οι ίδιες οι τράπεζες στις χώρες αυτές ε, αν είναι ο κύριος Παπαδόπουλος και εγώ δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος ε, ο δικαιούχος του λογαριασμού. Σε τέτοιες λοιπόν περιπτώσεις όταν δεν είναι σαφές σε ποιον ανήκει ο λογαριασμός δεν μπορεί κανείς να φέρει το βάρος απόδειξης. Ε, ε, νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε και τις διεθνείς αρχές να μπορούν να εντοπίζουν τους δικαίους των λογαριασμών. Εγώ έχω δει ε, και με την εμπειρία μου πιστεύω ότι αν κάποιος βλέπει ας πούμε ότι στο λογαριασμό Μόνικα Χολμάγε βρίσκονται 20 εκατομμύρια 200.000 αυτό είναι το πώς μπορεί κανείς να το εξηγήσει. Εγώ μπορώ ή δεν μπορώ να το κάνω. Ε, γι' αυτό συμφωνώ ε, ότι μπορεί να γίνει. Αλλά για λογαριασμούς τρίτων, ε, άγνωστους λογαριασμούς, ε, δεν νομίζω ότι είναι εύκολο να το κάνουμε αυτό. Δηλαδή είτε πρόκειται για κάποια περιουσιακά στοιχεία, για κάποιο λογαριασμό, θα πρέπει πραγματικός δικαιούχος να μπορεί να εντοπιστεί και να ταυτοποιηθεί, γιατί αλλιώς δημιουργούνται πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες της έρευνας και για τις αρχές αλλά και για τρίτους που δεν φταίνε και που δεν έχουν καμία σχέση Επομένως, ε, ε, πιστεύω ότι πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή τη γραμμή, την αυστηρή γραμμή του πραγματικού δικαιούχου, του beneficial owner, για να ξέρουμε ακριβώ σε ποιον ανήκει ο λογαριασμό και να διευκολύνουμε πολύ τη δουλειά στις αρχές. Ε, στη Γερμανία, παραδείγματο χάρη, υπάρχουν προβλήματα με κάποια οικόπεδα που δεν ξέρει κανεί ποιο είναι ο πραγματικό δικαιούχο και ποιο είναι αυτό που παίρνει το βάρος της απόδειξης. Το σύστημα του πόθεν έσχες ποιος είναι πραγματικός δικηγόρος είναι σημαντικό. Δεν ξέρω από πού, αν υπάρχει πίσω ένα δικηγορικό γραφείο κάποιος άλλος. Για μένα είναι πολύ σημαντικό να έχουμε την αρχή του πραγματικού δικαιούχου και για το ξέπλυμα χρήματο και για τη διευκόλυνση του έργου των αρχών. Έχω και προσωπική εμπειρία στον τομέα αυτό όπως είπα και τελικά είδα ε, ότι στην προκειμένη περίπτωση του δικού μας λογαριασμού ε, βρήκαμε τελικά ποιος ήταν ο δικαιούχος και τι ε, είχε γίνει με αυτά τα χρήματα. Δεν ήταν καθόλου ευχάριστο και σίγουρα καλό είναι τους απαταιώνες να τους ε, εντοπίζουν. Στην προκειμένη περίπτωση, ο δικός μας, το δικό μας το λογαριασμό που ήταν ανεργός και είχε χρησιμοποιηθεί από κάποιον άλλο, είναι πίσω από τα σίδερα ο απαταιώνας αυτός τώρα. Δεν το έψαξα σε ό,τι αφορά τα καλή opposed persons. Παραδείγματο χάρη έχουμε και κάποιου συμβολιογράφου, ε, ελεγκτέ που ασχολούνται με τον έλεγχο, ε, το audit ε, και κάνουν εκ μέρου του κράτου τέτοιου ελέγχου. Αυτό έχει τεράστια επίπτωση. Νομίζω ότι έχουν μεγάλη ευθύνη και αυτοί Άρα να μην συμπεριλάβουμε στην κατηγορία των, αυτών των ανθρώπων μόνο τους πολιτικούς ε, υπευθύνου, ε, αλλά και κάποιες άλλες κατηγορίες όπως αυτές που, που σας προανέφερα. Κάποιοι που μπορούν να πιστοποιούν ε, τα βιβλία, τα λογιστικά ή τους λογαριασμούς, παραδείγματος χάρη μπορεί να έχουν εμπλακεί σε τέτοιες δραστηριότητες ξεπλήματο ε, ή μπορεί να μην φταίνει και να τους ε, εμπλέξουν σε τέτοιες δραστηριότητες. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήταν καλό να ακούσουμε για αυτό το τεκμήριο αθωότητας ε, την άποψη του εισηγητού, γιατί υπάρχει και οδηγία της κύρια Γκρισμπέκ. Το τεκμήριο αθωότητας δεν ξέρω αν αυτά τα δύο συνδέονται. Εγώ καταλαβαίνω τι εννοείται, αλλά θα μας πει η συγγήτρια και τη δική της άποψη, μάλλον η και τη δική του άποψη. Τώρα, η Άννα Γκόμης εκ μέρους των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Σας ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ με τη Μόνικα. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τις συζητήσεις που είχαμε, κατά τις οποίες καταφέραμε να κάνουμε πολλή δουλειά προσπάθησε να συγκεράσει τις διάφορες απόψεις για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Θα ήθελα να επικεντρωθώ στα σημαντικά για μένα στοιχεία και για τα οποία έχω υποβάλει τροπολογίες. Φορολογικά εγκλήματα. Θεωρούνται κύρια εγκλήματα στην predicate offenses, στην ε, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, ε, η διατύπωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όμως ε, αφήνει μεγάλο περιθώριο ευελιξίας, ε, μεγάλο περιθώριο διακριτικής ευχέρειας στα κράτη-μέλη. Ε, αυτό το περιθώριο διακριτικής ευχέρειας εμείς θέλουμε να το περιορίσουμε. Άσχετα από τα κατόφλια που υπάρχουν στην εθνική νομοθεσία. Όσον αφορά τις, την φοροδιαφυγή και τέτοια. Για να είναι αποτελεσματική η νομοθεσία κατά της ε, νομοποίησης παράνομων εσόδων, ε, δεν ε, θα πρέπει να είναι απαραίτητο να καθορίσουμε το έγκλημα που έχει οδηγήσει στα παράνομα έσοδα, πόσο μάλλον να υπάρξει καταδίκη. Επίσης, δεν θα πρέπει να εμποδίζεται η καταπολέμηση το, τις ε, παράνομων εσόδων ε, από το αν έχει πραγματοποιηθεί το κύριο έγκλημα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε, ή τρίτη χώρα. Άσχετα λοιπόν από το αν το κύριο έγκλημα θεωρείται έγκλημα στο, στη δικαιοδοσία όπου πραγματοποιήθηκε και μιλάμε για ε, εμπόριο ναρκωτικών, για εμπορία ανθρώπων κλπ. Επίσης, η δυνατότητα των κρατών μελών ε, να ποινικοποιούν ε, πράξεις που δεν συμπεριλαμβάνονται στην αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για να διασφαλίσω την αναλογικότητα, ε, έχουμε συμπεριλάβει την αμέλεια ως κύριο έγκλημα για νομικά πρόσωπα, σαν νομικά πρόσωπα γνωρίζουμε τους κινδύνους στον ε, αγώνα της καταπολέμησης ε, της νομοποίησης παράνομων εσόδων ε, και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ποινικοποιούν την αμέλεια όταν με βάση τα στοιχεία είναι σαφές ότι ο ύποπτος θα έπρεπε να γνωρίζει ότι τα έσοδα αυτά προέρχονται από κλιματικές δραστηριότητες. Τέλος, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει εάν σύμφωνα με την οδηγία αυτή είναι κανείς υπόχρεος ή αν έχει διαπράξει έγκλημα στο πλαίσιο μιας εγκληματικής οργάνωσης, αυτό θα αποτελεί επιβαρυντικό παράγοντα. Επίσης προσθέτω ότι εάν μιλάμε για πολιτικά εκτεθειμένο πρόσωπο και αυτό θα πρέπει να είναι επιβαρυντικό στοιχείο και στο θέμα αυτό συμφωνώ με αυτά που υπόθηκαν από συναδέλφους σχετικά με τις ελάχιστες ποινές. Έχω εισάγει και την αρχή των ελάχιστων ποινών φυλάκισης για ε, τους εγκληματίες όταν υπάρχουν και αυτά τα επιβαρυντικά στοιχεία. Ευχαριστώ πολύ. Η Μόνικα Μακοβέη είναι σκιώδης συγγήτρια για το ECR. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Ιγνάτσιο για όλες τις προσπάθειές του και για τις εξαιρετικές προτάσεις που έχει υποβάλει. Να ευχαριστήσω και τους ε, συναδέρφους ε, που υπέβαλαν παρόμοιες τροπολογίες. Κάποιες από αυτές που να οδηγήσουν σε μεγάλες συζητήσεις. Είμαι βέβαιη όμως ότι θα καταλήξουμε σε συμβασμό. Οι δικές μου τροπολογίες έχουν να κάνουν με το εξή. Πρέπει να έχουμε την ευκαιρία να καταδικάζουμε εγκληματικές πράξεις ε, ακόμη και αν το πρόσωπο δεν έχει καταδικαστεί για την ε, εγκληματική πράξη που οδήγησε στα παράνομα έσοδα. Πιστεύω λοιπόν ότι η νομοποίηση παράνομων εσόδων ε, θα πρέπει να αρκεί από μόνη της για κατάσχεση και δίμευση. Το πρόβλημα δηλαδή εδώ είναι η έλλειψη κυρίου εγκλήματος. Εάν το πρόσωπο αυτό είναι ένοχο διαφθοράς και ε, νομιμοποιεί τα παράνομα έσοδα από ε, τη διαφθορά, δεν, ε, αυτό θα πρέπει να αρκεί από μόνο του. Επίσης, οι παράνομες πηγές εσόδων που ξεπερνούν το νόμιμο εισόδημα. Ο ένοχος δηλαδή θα πρέπει να αποδείξει ότι η πηγή του πλούτου του είναι νόμιμη εφόσον ξεπερνά το νόμιμο του εισόδημα. Θα διαφωνήσω με την κυρία Χολμάγερ όσον αφορά το βάρος της απόδειξης. Εάν κάποιος έχει ένα εκατομμύριο ευρώ νόμιμο εισόδημα και τα περιουσιακά του στοιχεία ανέρχονται σε δέκα εκατομμύρια, εδώ δεν μιλάμε για αντιστροφή του βάρους της απόδειξης, μιλάμε για την νόμιμη υπεράσπιση. Ο δικαστής θα ζητήσει από τον εισογγελέα να αποδείξει ποια είναι τα περιουσιακά στοιχεία του προσώπου και ποιο είναι το νόμιμο εισόδημα του προσώπου αυτού. Εάν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στα δύο αυτά, ε, το πρόσωπο, ο ε, ύποπτος θα πρέπει να αποδείξει από πού προέρχονται τα στοιχεία αυτά. Όταν κάποιος κατηγορείται για έγκλημα, θα πρέπει να αποδείξει ότι είναι αθώος. Ε, γι' αυτό λοιπόν είμαι υπέρ ε, του να πρέπει να αποδείξει κανείς ε, από πού προέρχεται από πού προέρχονται τα περιουσιακά του στοιχεία. Επίσης, έχουμε Ε, περιπτώσεις ύποπτων ε, μεταφορών μετρητών μέσω τρίτων για να είναι δύσκολη η ανείχνευση. Στην πέμπτη οδηγία για την καταπολέμηση της νομοποίησης παράνομων εσόδων ε, θέλουμε να εμποδίσουμε κάποιες πράξεις ώστε να μπορέσουμε να εντοπίσουμε τις περιπτώσεις αυτές. Και στην οδηγία αυτή θέλουμε να συμπεριλαμβάνεται ακριβά το ίδιο, διότι είναι πολύ δύσκολο να απαγορεύσει κανείς τέτοιες πράξεις. Απαγορεύονται σε κάποια κρατημέλη, υπάρχουν περιορισμοί σε άλλα κρατημέλη. Στη Ρουμανία όμως δεν υπάρχει κανένας περιορισμός. Θα ήθελα να σας θυμίσω ότι εδώ μιλάμε για ανώνυμα έγγραφα Ε, είναι δηλαδή κανείς ε, ιδιοκτήτης των μετόχων σε μια εταιρεία εφόσον έχει αυτό το χαρτί στη τσέπη του. Δίνει το χαρτί σε κάποιον άλλον, είναι πια άλλος ο ιδιοκτήτης, ο κάτοχος. Ε, κανείς λοιπόν ε, δεν γνωρίζει ποιος είναι ο νόμιμος δικαιούχος ή ιδιοκτήτης των μετοχών αυτών Αυτέ τι μετοχέ, ε, λοιπόν μπορείς να τη διαβιβάσει κανείς ε, χωρίς καμία δυσκολία. Δεν έχουν ε, θέση όμως στο πλαίσιο τη καταπολέμησης της απάτης. Δυστυχώς ο κυβερνοχώρος δεν ρυθμίζεται. Έχουμε ε, εικονικά νομίσματα, bitcoins, κρυπτονομίσματα, κυβερνοεπιθέσεις, ιούς στους υπολογιστές με τους οποίους ζητείτε, ζητούνται λίτρα για να πάρει κανείς πίσω τα δεδομένα του. Με τις τροπολογίες μας λοιπόν ζητάμε εργαλεία ώστε αυτοί που διερευνούν το κυβερνοέγκλημα να είναι σε θέση να τα καταπολεμήσουν αυτά τα φαινόμενα. Τέλος, Θέλουμε πιο αυστηρές ποινές για πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα. Σε αυτό συμφωνούμε όλοι και θέλουμε συμπληρωματικές ποινές για πρόσωπα και επιχειρήσεις που νομιμοποιούν έσοδα από παράνομες δραστηριότητες. Πολιτικοί λοιπόν που έχουν παραπάνω ευθύνη μπορεί να βρίσκονται στην εξουσία ή όχι. Όταν όμως βρίσκονται στην εξουσία έχουν πρόσβαση σε διάφορους πόρους, γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχουν περισσότεροι περιορισμοί για πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα, όταν για παράδειγμα ανοίγουν ένα λογαριασμό. Και θα πρέπει οι ποινές να είναι πιο αυστηρές σε περίπτωση εγκλήματος. Πρόσθετες ποινές, ε, ε, πρόσθετες ποινές λοιπόν ε, απαγόρευση ε, συμμετοχής σε δημόσιες ε, συμβάσεις και μιλάμε για δημάρχους, υπουργούς κλπ. Καμία πρόσβαση σε δημόσιες ε, θέσεις, σε δημόσια αξιώματα. Αυτές λοιπόν είναι πρόσθετες ποινές για τα πρόσωπα αυτά. Θα κλείσω εδώ. Προσλέπω στην επόμενη εβδομάδα στις ε, δύο συναντήσεις που θα έχουμε με τους ε, ε, διάφορους σκιώδεις συζητητές. Ευχαριστώ πολύ. Μόνικα, θες να επανέλθεις σύντομα. Αγαπητοί συνάδελφοι, Όσον αφορά αυτό που είπε η Μόνικα, έχω την ε, εντύπωση ότι διάφορες ε, οδηγίες δεν έχουν εφαρμοστεί σωστά. Ανώνυμοι τραπεζικοί λογαριασμοί εδώ και πολύ καιρό δεν επιτρέπεται να υπάρχουν. Ε, νωρίτερα στην Αυστρία αυτό συνηθιζόταν και σε άλλα κράτη-μέλη. Όπου στο όνομα γράφεται Χ. Αλλά αυτό εδώ και πολύ καιρό απαγορεύεται. Αυτό που δεν απαγορεύεται είναι ο πραγματικό δικαιούχο να είναι άλλο. Και αυτό το βλέπουμε στην Ειδική Επιτροπή για τα έγγραφα του Παναμά, όπου ο ιδιοκτήτης κρύβεται πίσω από κάποια άλλη δομή. Μόλις αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα θα γνωρίζουμε ποιος είναι ακριβώς ο πραγματικός δικαιούχος ε, ενός τραπεζικού λογαριασμού, μιας επιχειρήσης κλπ. Γι' αυτό το θέμα του πραγματικού δικαιούχου είναι πολύ σημαντικό. Οι αρχές θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές και μιλώ και για τις φορολογικές αρχές και για τους εισαγγελείς. Ε, επίσης υπάρχουν οι εκθέσεις για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης παράνομων των τραπεζών. Θα πρέπει λοιπόν υπάρχει η δυνατότητα να εντοπιστεί ο πραγματικός δικαιούχος ε, και να διερευνηθεί. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε συστηματικές δομές που να διασφαλίζουν κάτι τέτοιο. Και θα πρέπει να εφαρμόζεται σωστά η οδηγία σε όλα τα κράτη-μέλη. Βλέπουμε λοιπόν ότι η οδηγία δεν εφαρμόζεται ε, επαρκώς ε, σε κάποια κράτη-μέλη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να υποβάλει πάρα πολύ ωραίε προτάσει, αλλά διαπιστώνουμε ότι στη Ρουμανία, για παράδειγμα, συνεχίζει να είναι δυνατόν ε, να μπορεί κανεί να έχει ανώνυμο τραπεζικό λογαριασμό. Αυτό όμω απαγορεύεται εδώ και πολύ καιρό. Και ο πραγματικό δικαιούχο είναι ένα κενό, ένα παραθυράκι το οποίο θα πρέπει να κλείσουμε, διότι είναι κάτι που εκμεταλλεύονται οι εγκληματίες και τους δίνει εξαιρετικές δυνατότητες για να κρύψουν την, ε, ταυτότητά τους. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, Μόνικα. Εγώ αυτό που θέλω ε, είναι να εφαρμοστούν οδηγίες αυτές. Στο Κοινοβούλιο, για παράδειγμα, στη Ρουμανία, έχουμε τώρα την ε, τέταρτη οδηγία κατά του ξεπλήματος χρήματος. Τέσσερα κράτη, Ισπανία, Πορτογαλία, Ρουμανία και ένα άλλο είναι τα τέσσερα κράτη-μέλη που δεν υπάρχουν ε, όρια. Παραδείγματο χάρη για αυτές τις ε, μετοχές ε, που γράφουν στον κομιστή. Και είναι μάχη το να μπορέσουμε να έχουμε πρόσβαση στους πραγματικούς δικαιούχους των εταιριών και εγώ προσπαθώ δεξιά αριστερά, από εδώ από εκεί δεν ε, ξέρω τι κάνει η κυβέρνησή μας, γιατί δεν μεταφέρει αυτή την οδηγία. Δεν ξέρω μήπως ε, φοβούνται. Ωραία, τώρα θέλει και Άννα το λόγο, λέει ο Πρόεδρος. Ναι, εγώ θέλω να πω συμφωνώ με τη Μονικά να διορθώσω. Η χώρα μου, η Πορτογαλία, μόνος, ε, μόλις απαγόρεσε αυτές τις του είδους τις μετοχές στον κομιστή και τους αναγκάζει να καταγράφουν τον ε, πραγματικό δικαιούχο. Βρίσκουν βέβαια τρόπους ε, πολύ ενδιαφέροντες για να παρακάμψουν. Βλέπω ότι σας μαθαίνουν ε, οι σκιώδεις τηγέτες στις χώρες τους, σε πράγματα που αυτή είναι, αυτή είναι η αξία αυτών των συζητήσεων εδώ και ο πλούτος των συζητήσεων. Σας ενημερώνουν λοιπόν για το τι γίνεται στις χώρες τους οι συνάδελφοι. Κύριε Κοράου, να ακούσουμε σύντομα την Κομισιόν, πες σας δώσω ξανά το λόγο. Ή και και Κατερίνα μήπως. Σίγουρα. Γιατί περίμενες υπομονετικά Κατερίνα. Όχι, δυστυχώς πρέπει να φύγω. Την επόμενη φορά θα σας πω. Ευχαριστώ που παρακολούθησε τη συζήτηση. Ξέρω ότι ενδιαφέρεσαι για αυτό το θέμα. Δύο λόγια να ακούσουμε και από την Επιτροπή γρήγορα γρήγορα. Λίγη υπομονή κύριε Σιγητά. Ευχαριστώ. 182 τροπολογίες. Πρέπει να σας πω ότι είμαστε αισιόδοξοι. Και γιατί τα βασικά σημεία δεν τα έχετε πειράξει, από την πρόταση της Κομισιόν, αλλά και επίσης αυτά που προτείνεται ως ΛΥΜΠΕ θεωρούμε ότι είναι και πολύ καλά. Υπάρχουν πολλές τροπολογίες ε, που μπορούν να αυξάνουν τα αποτρεπτικά μέσα, δηλαδή αύξηση των ποινών κτλ. Άλλες τροπολογίες μπορούν να βελτιώσουν τη συνεργασία περιορίζοντας ε, τους όρους ε, για τις διώξεις και τις έρευνες, το είπε και ο εισηγητής του Επικιάνα Γκόμες. Μιλάμε για την περίπτωση χάρη, όπου οι πρόσοδοι φτάνουν σε άλλη χώρα από εκεί έχει το ξέπλυμα και η αρχική πρόταση της Κομισιόν λέει ότι μπορεί να περιοριστούν οι διαδικασίες στην περίπτωση που το ποινικό αδίκημα έχει γίνει εκτός. Έχουμε όμως και θέματα όπως είναι η πειρατεία, διαφθορά, διακίνηση ανθρώπων, σεξουαλική εκμετάλλευση. Υπάρχουν παραθυράκια στις τρίτες χώρες και είναι δύσκολο να πούμε ότι με διερεύνηση, ε, μάλλον ότι αυτές οι δραστηριότητες θα παραμείνουν ατιμόρυτες. Υπάρχουν και διαφορετικοί κανόνε, πάνω χάρη για τι αμβλώσει, τα ναρκωτικά και την ευθανασία. Δεν ξέρω αν πρέπει ε, να επιλέξουμε την προσέγγιση του εισηγητού και τροπολογία Κινίτσι Γκόμες. Τρία σχόλια ακόμη θέλω να κάνω. Το πρώτο, ένα από του βασικού μα στόχου είναι να είναι ευρύ αρκετά το πεδίο εφαρμογή για να καλύπτονται οι πρόσοδοι από όλε τι εγκληματικέ δραστηριότητε σημαντικέ, δηλαδή και τι φορολογικέ. Εσεί θέλετε να υπάρχει ένας πιο εξέχων ρόλος και θα το δούμε. Για το ξέπλυμα χρήματος. Στις περισσότερες περιπτώσεις το κάνουν οι ίδιοι εγκληματίες και δεν ξέρω, με κάποιες τροπολογίες νομίζω ότι τορπιλίζονται οι στόχοι μας και το άλλο. Πριν καταδικαστεί κάποιος για ξέπλυμα χρήματος. Υπάρχουν κάποιες προτάσεις ε, που δεν θα επιτρέψουν ε, την ε, σωστή αντιμετώπιση του ζητήματος από την ποινική δικαιοσύνη. Θα τα δούμε αυτά, επιμένω και την ψηφοφορία στις 13 Νοεμβρίου. Ωραία. Με όλα αυτά φτάσαμε στο τέλος, δίνω το λόγο στον Ιγνάσιο. Σας ευχαριστώ. Τώρα χαίρομαι που άναψε η συζήτηση, ακόμα και αν ε, ίσως να βγει και πέρα από το θέμα αυτής της ε, οδηγίας. Πάντως είναι σίγουρα πάντα ενδιαφέρον μέσα σε μια κοινοβουλευτική ε, ε, επιτροπή να γίνει συζήτηση. Τώρα, όσον αφορά το βάρος της απόδειξης, ήθελα να και το είπε και η Μόνικα Ολμάγερ, Τη λογική λοιπόν για το βάρος της απόδειξης θα πρέπει να επαναλάβουμε ότι σε οποιοδήποτε σύστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως και στο Ιταλικό η αντιστροφή του βάρους της απόδειξης δεν αφορά την, ε, το ίδιο το ποινικό αδίκημα, αλλά το μέτρο της ε, ε, περιουσίας, δηλαδή σχετίζεται με την κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων που είναι αναμονή. Δηλαδή είναι μια ένα προληπτικό μέτρο, δεν είναι ποινή. Δεν είναι... μπορεί να επεκταθεί δηλαδή και στην αντίστροφή του βάρους απόδεξης. Τώρα, μιλήσατε για συμβολογράφους, για αυτούς που στο εσωτερικό ενός συστήματος χαίρουν μιας εμπιστοσύνης. Υπάρχει το ε, σε το άρθρο 6β που αναφέρεται σε αυτό το είδος τους ανθρώπους ως ε, επιβαρυντική περίσταση. Νομίζω πως ήδη υπάρχει αυτό δηλαδή. Ε, δεν ξέρω αν αυτή ήταν η ερώτηση ή αν έπρεπε να διατηρηθεί αυτό το είδος η προσέγγιση. Πάντως πιστεύω πως αυτή η προσέγγιση είναι σωστή. Ότι δηλαδή είναι επιβαρυντικό στοιχείο το όταν κανείς έχει ένα ιδιαίτερο δημόσιο αξίωμα όσον αφορά την Άννα Γκόμες που αναφέρθηκε στο στα φορολογικά δικήματα, δηλαδή το γεγονός ότι η φοροδιαφυγή θεωρείται πάντοτε ως ε, αδίκημα. Εδώ υπάρχει πρόβλημα εναρμόνισης των φορολογικών αδικημάτων, των αδικημάτων φοροδιαφυγής. Το ίδιο πράγμα, το ίδιο είδος αδικήματος δεν θεωρείται το ίδιο ανάλογα με το σύστημα του κάθε κράτους μέλους της Ένωσης. Η φοροδιαφυγή για 1000 ευρώ μπορεί να θεωρηθεί αδίκημα κάπου, ενώ αλλού όχι. Πριν να φτάσουμε λοιπόν στην ε, ορισμό ενός ε, αδικήματος ε, θα πρέπει να έχουμε μια βοήθεια από πλευράς της Επιτροπής για την εναρμόνιση του ορισμού του, του, του, του αδικήματος της φοροδιαφυγής σε ολόκληρη την Ένωση για να... θα ήταν σωστό αυτό για να μην έχουμε όλα αυτά τα προβλήματα που τώρα αντιμετωπίζουμε ε, με, το, ότι με, αυτούς που μετακινούνται ας πούμε για να έχουν πιο ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση από κράτος σε κράτος, αλλά έτσι με μια ολόκληρη πολιτική συζήτηση. Ε, για τα κατά τα λοιπά πιστεύω πως ε, πολλές παρατηρήσεις ε, με βρίσκουν σύμφωνο. Θεωρώ ότι θα είναι καλή ευκαιρία να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα και να βρούμε και σημεία επαφής. Και σας ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σας και για τις τροπολογίες που υποβάλατε. Αυτά. Χριστό Γινάσιο και καλή επιτυχία με τις ε, συνεδριάσεις των ε, σκιωδών. Σας ευχαριστώ που ήρθατε πέμπτη απόγευμα και για τον πλούτο αυτής της συζήτησης. Η ψηφοφορία προβλέπεται για τις 13 Νοεμβρίου. Κλείνουμε έτσι και φτάνουμε στα διάφορα. Ε, αν δεν υπάρχει τίποτα στα διάφορα, είναι το τέλος της συνεδρίασης. Η επόμενή μας συνεδρίαση είναι για τις 6 Νοεμβρίου. Ευχαριστώ συνάδελφοι.